die wissen das. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Σήμερα κάνουμε μια ακρόαση για να δούμε μετά από ένα χρόνο τη δουλειά της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, πώς έχουν οι εξελίξεις, πόσο έχει η συνεργασία μεταξύ της υπηρεσίας και της Κομισιόν και κάποια άλλα πράγματα και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι στην πρώτη συζήτηση έχουμε τόσους ικανούς εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων και του ελεγκτικού συνεδρίου βλέπουμε πως το 2013 θα έχουμε μια αναθεώρηση και πρέπει να προετοιμαστούμε αναλόγως εξού και η σημερινή ακρόαση οπότε δεν θα έχουμε σχέδιο ψηφίσματος μετά από αυτή την ακρόαση δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά ε, απλά ως διαδικασία. Είναι μέρος μιας διαδικασίας διαρκούς για το πώς θα διαμορφωθούν το κοινού πολιτικές σχετικές. Χαίρομαι για το ότι είχε έρθει και ο Επίτροπος ο κ. Σεύκοβιτς και η Γενική Γραμματέας η Κάθριν Τζέι. Χαίρομαι επίσης για το ότι έχουμε κορυφαίο στελέχη της υπηρεσίας αυτής, ο Πιέρ Μπεμό και ο κύριος ο Σάλιβαν και χαίρομαι επίσης για το ότι και ο κύριος Πίνξτεν είναι εδώ πέρα, μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. καθηγητής του Πανεπιστημίου της Λουβέν και του Κολεγίου της Ευρώπης. Υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία και θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στους για πέντε λεπτά να κάνουν μια αρχική δήλωση και ελπίζω οι δύο αυτές ώρες να χρησιμοποιηθούν με τρόπο σωστό. Λοιπόν, δεν θα καθαρίσω άλλο, μπορούμε να περάσουμε μέσω στην συζήτηση. Πρώτα απ' όλα τον λόγο έχει ο κύριος Επιτροπός, ο κύριος Σεύκοβιτς. Thank you uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και εσάς προσωπικά για την ιδέα που είχατε να διοργανώσετε την ανταλλαγή απόψεων για την πρόοδο που σημειώσαμε μετά την σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Χαίρομαι επίσης που Έχουμε εδώ και τον Γενικό Εκτελεστικό Γραμματέα, τον κύριο Βημόν, τον Διοικητικό, το Διοικητικό Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Σάλιβαν και πολύ στενούς συνεργάτες της κυρίας Κάθη Έξτον που θα μας μιλήσουν για το πώς έχει επιτελέσει το έργο της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ήταν καταπληκτική συνεργασία που είχαμε τα τελευταία διετία και από πρακτική και από πολιτική άποψη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερική Δράση. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι φαίνονται οι καρποί αυτή τη συνεργασία. Η απόκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αραβική Άνοιξη με κοινή ε, με κοινέ στρατηγικές που συνδυάζουν την ΚΕΠΑ και τι δραστηριότητε και αρμοδιότητες Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επίση, τα έγγραφα προγραμματισμού Εξωτερική αρρωγή και αγαστή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι προτάσει ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου για τα εξωτερικά μέσα και μηχανισμού που έχετε λάβει. Τώρα από κοινό προετοιμάζουμε τις διασκέψεις κορυφής με τρίτες χώρες με τους Προέδρους Μπαρόζο και Βανερόν Πόη, το Ευρωπαϊκό Έργο για τις Κυρώσεις, προετοιμασία και διεξαγωγή διεθνών διαπραγματεύσεων με διεθνείς εταίρους, ενώ ανέκαθεν φυσικά σεβόμασταν τις αρμοδιότητες του ενός και του άλλου οργάνου. Έχουμε καθημερινή συνεργασία επιτόπου στις αντιπροσωπείες ε, με συνεργασία του προσωπικού της ΕΕΔ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα συλλογικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπό την αιγύδα φυσικά του επικεφαλής αντιπροσωπείας προγραμματίζοντας και εξασφαλίζοντας μια συνέχεια των προγραμμάτων συνδρομής ή διαμηνύοντας ε, τις πολιτικές, για παράδειγμα, τις ε, συμμαχίες ε, που προσπαθούμε να διαμορφώσουμε εν ώψη της διάσκεψης του Ντέρμπαν. Φυσικά υπήρχαν κάποιες δυσκολίες τα πρώτα δύο χρόνια στο ροντάρισμα και αυτό ήταν απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μιας νέας πραγματικότητας μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας προκειμένου να εφαρμόσουμε την απόφαση για την ΕΙΕΔ εντός του θεσμικού πλαισίου και των θεσμικών κανόνων. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι οι αναμενόμενες αυτές προκλήσεις αντιμετωπίστηκαν με πολύ επικοδομητική συνεργασία. Για παράδειγμα, μερικά διοικητικά θέματα που χαρακτηρίστηκαν ως εκρεμή στις, στην έκθεση της είπαν εκπροσώπου στα τέλη Σεπτεμβρίου ήδη είχαν επιληθεί τις πρώτες εβδομάδες του τρέχοντος έτους και οι απαραίτητες ρυθμίσεις και κατευθυντήριες γραμμές στόχο έχουν να καθοδηγήσουν και τους αξιωματούχους και τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών. Όλοι γνωρίζουν στο επίπεδό τους τι θα πρέπει να κάνουν και με ποιο τρόπο. Έτσι εξασφαλίζεται ε, η ομαλή διεξαγωγή ε, του έργου της κάθε αντιπροσωπείας και επίσης έχουμε δώσει και εσωτερικές οδηγίες στο προσωπικό για να συνεχιστεί η συνεργασία με τους συναδέλφους της ΕΙΕΔ στέλνοντας οδηγίες ε, ή πληροφορίες στις διάφορες αντιπροσωπείες. Για παράδειγμα, κοινέ οδηγίε τη ΕΕΔ και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεστάλησαν σε όλου του επικεφαλεί αντιπροσωπιών στι 20 Δεκεμβρίου, διευκρινίζοντα ε, τα καθήκοντα κάθε κατηγορία ε, υπαλλήλου των αντιπροσωπιών. Οι οδηγίε καλύπτουν ε, πρώτα αρχικά καθήκοντα και βασικά καθήκοντα του κάθε υπαλλήλου στην αντιπροσωπεία, η απαραίτητη ελαστικότητα που θα πρέπει να επαφίεται και το περιθώριο λιγμών στον επικεφαλής αντιπροσωπείας, προκειμένου η αντιπροσωπεία να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις της και στο φόρτο εργασιών, φυσικά ε, με σεβασμό των νομικών απαιτήσεων του δημοσιονομικού κανονισμού και του υπηρεσιακού κανονισμού. Πρόσφατα συμφωνήσαμε και σε κάποιους κανονισμούς για να συντονίσουμε τη διαχείριση του προσωπικού μας αντιπροσωπείας, αντικαθιστώντας προηγούμενους μηχανισμούς που ίσχυαν εντό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεδομένου του ρόλου που θέλουμε να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο, θέλουμε ε, τακτικά να αναθεωρούμε τα επίπεδα του προσωπικού και να ε, αφιερώνουμε το προσωπικό στα καθήκοντα που είναι τα πιο απαραίτητα και στις περισσότερες, μεγαλύτερες προτεραιότητες. Γι' αυτό θα, θα αποσπάσουμε τους υπαλλήλους μας ανάλογα με τις προτεραιότητές μας. Θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα κριτήρια για να δούμε πόσοι πάλι χρειάζονται πού, ανάλογα με, το, με τα κονδύλια που έχουμε φυσικά στις διάφορες αντιπροσωπείες και θα αξιολογήσουμε και, τις και το κατά πόσο είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε την παρουσία μας σε κάποιες βασικές αντιπροσωπείες για βασικούς τομείς όπως είναι η ενέργεια, το περιβάλλον και οι εσωτερικές υποθέσεις. Μια και θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις, ε, τη μείωση κατά 5% του προσωπικού, προτείναμε στην αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή να ε, στελεχώσουμε τις αντιπροσωπείες ε, σταδιακά και για μια σειρά ετών. Θα ήθελα εν κατακλείδη να επαναλάβω την συνεχή υποστήριξή μας και την αμύωτη υποστήριξη και συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε όλα τα επίπεδα, εξασφαλίζοντας ομαλή συνεργασία μεταξύ όλων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλές επαφές με τους συναδελφούς της ΕΙΕΔ κοινό μα στόχο είναι η προγωγή των συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαδραματίσουμε το στρατηγικό ρόλο που περιμένουν όλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε τώρα με ποιο τρόπο θα πρέπει να συνεργαστούμε, γιατί έχουμε λύσει τι ε, βασικές, αρχικές μας και πιστεύω ότι με τι κοινέ προσπάθειε θα έχουμε πραγματικά ε, προσεθέμενη αξία και σημαντική διαφορά. Ο κύριο Βημό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια. Θα πρέπει να σας πω ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και αισθανόμαστε μεγάλη, μας κάνετε μεγάλη τιμή που μας καλέσατε σήμερα εδώ μαζί με τον David. Θα πρέπει να σας πω ε, ποια είναι η εργασία που κάνουμε στην ΕΕΔ για τα τελευταία δύο χρόνια περίπου. Το πρώτο έτος βασικά ε, έπρεπε να στήσουμε τις νέες υπηρεσίες ε, κατά κάποιο τρόπο προσγειωθήκαμε και αμέσως έπρεπε να αρχίσουμε να τρέχουμε γιατί είχαμε άμεσα κρίσεις να αντιμετωπίσουμε στη διεθνή κοινότητα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησε η ΕΕΔ ήταν ε, η κρίση που ξεκίνησε στην Λευκορωσία μετά τις προεδρικές εκλογές και έπειτα συνεχίσαμε με ένα σωρό διαφορετικά γεγονότα στον αραβικό κόσμο, αυτό το οποίο τελικά ονομάστηκε Αραβική Άνοιξη. Αν θέλουμε να συνοψίσουμε, βασικά κάναμε τρία πράγματα. Το πρώτο ήταν να φτιάξουμε και να εφαρμόσουμε τις νέες ευρωπαϊκές ε, αντιπροσωπείες και να ορίσουμε το είδος συνεργασίας που θέλουμε να κάνουμε με τα κράτη-μέλη επί τόπου. Έχουμε φτιάξει κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με το είδος συνεργασίας και καλής πρακτικής που θέλουμε να προωθήσουμε Επίσης, θεσπίσαμε κατευθυντήριες γραμμές για τις διάφορα, τα διάφορα διπλωματικά διαβήματα και την ανταλλαγή πληροφοριών και μέχρι στιγμή η εντύπωση που έχουμε και η υποδοχή που είχαμε από πλευρά των κρατών είναι ότι όλα βαίνουν καλώς. Το δεύτερο είναι ότι θελήσαμε να φτιάξουμε τον μέθοδο εργασίας μας εδώ στις Βρυξέλλες, στο Γενικό Επιτελείο και το Συμβούλιο και ο ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος ανέλαβαν το, με την ε, περιτροπή της Προεδρίας είτε μέσω των διαφορών ομάδων εργασίας είτε διάφορα συμβούλια εξωτερικών υποθέσεων ή ανάπτυξης Έπρεπε να φτιάξουμε και τις σχέσεις μας, να ορίσουμε τις σχέσεις μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το πολιτικό θέμα της πολιτικής ε, λογοδοσίας τρίτο έργο ήταν να να εφαρμόσουμε νέους τρόπους εργασίας, νέες πρακτικές σε όσα σχετίζονται με τη διαχείριση κρίσεων. Ε, φτιάξαμε δημιουργήσαμε ένα νέο στυλ εργασίας στην ΕΙΔ με την ε, πλατφόρμα κρίσης, με τη συγκέντρωση όλων όταν αντιμετωπίζουμε κρίση όπως στη Συρία ή στη Λιβύη ή αλλού. Και νομίζω ότι από όσο μπορούμε να δούμε μέχρι στιγμής, σίγουρα Όλα αυτά θα πάρουν καιρό, αλλά μέχρι στιγμής ξεκινήσαμε καλά και προχωράμε καλά. Αν δούμε το δεύτερο έτος λειτουργίας της ΕΕΔ, ε, νομίζω πως τώρα θα πρέπει να σταθεροποιήσουμε τα όσα κάναμε τον πρώτο χρόνο. Θα έλεγα ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρεις κεντρικές προκλήσεις. Η πρώτη αφορά την ε, οικοδόμηση μιας νέας διοικητικής κουλτούρας. Έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Αυτό σημαίνει βελτίωση του τρόπου συνεργασίας μας, να ε, συνεργάζονται δηλαδή όλα τα διάφορα στοιχεία της υπηρεσίας προς την ίδια κατεύθυνση. Δεύτερον, να αναλαμβάνουμε περισσότερες πρωτοβουλίες γιατί τα κράτη-μέλη ζητούν πνευματική, όπως την λένε, ε, ε, ηγετική πρωτοβουλία. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε. Και έπειτα θέλουμε να μπορούμε να ενεργήσουμε πιο γρήγορα. Έτσι όπως είναι οργανωμένο το σύστημα, παίρνει χρόνο η λήψη αποφάσεων και η εφαρμογή των δράσεων με σωστό τρόπο. Όταν αντιμετωπίζουμε γεγονότα σε εξέλιξη όπως στην Λιβύη, τη Συρία, είναι αναγκαίο να είμαστε επιτόπου γρήγορα, να είμαστε ταχύτεροι στις αντιδράσεις μας και να ε, μπορούμε να εφεύρουμε νέους τρόπους μαζί με την Κομισιόν και τα κρατημέλη για να ενεργούμε πιο γρήγορα. Η δεύτερη πρόκληση είναι αυτή η περίφημη ολοκληρωμένη προσέγγιση. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με ολοκληρωμένη προσέγγιση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, όχι μόνο να χρησιμοποιήσουμε τα συνηθισμένα διπλωματικά μέσα, αλλά να εκμεταλλευτούμε και όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και τέλος έλεγα και ξέρω πως αυτό είναι ιδιαίτερα προσφυλές για πολλούς ευρωβουλευτές, αφορά τη στρατηγική και το στρατηγικό όραμα. Και εδώ χρειάζεται να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε και να έχουμε περισσότερη στρατηγική ε, στρατηγικό όραμα. Ε, δεν ε, μιλάμε μόνο για ευρωπαϊκή στρατηγική. Τα περισσότερα μέλη μας είπαν ότι θέλαν κάτι λιγότερο φιλόδοξο, αλλά κάτι που το οποίο στην ουσία θα ιεραρχεί τις σωστές προτεραιότητες, θα προγραμματίζει τις δράσεις για τα επόμενα χρόνια, ώστε να έχουμε έναν γνώμονα για το που θέλουμε να φτάσουμε. Αυτά έχω να πω και να, αφήσω το, να δώσω το λόγο ίσως στον David. Ευχαριστώ πολύ, Πιέρ, ο David. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αν μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως ο στόχος της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης είναι η πολιτική και η παραγωγή αυτής, είναι γεγονός πως ε, το πρώτο έτος μεγάλη πρόκληση ήταν μόνο και μόνο να οργανωθούμε. Ε, μόνο η δικιά μας διοίκηση ε, ασχολείται περισσότερο με την οργάνωσή της παρά με την παραγωγή έργου, αλλά είναι, ήταν νέος ο οργανισμός ε, και αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι έπρεπε να συναρμολογήσουμε ένα έπιπλο χωρίς οδηγίες και δεν ξέραμε αν είχαμε και όλα τα κομμάτια. Οι πρώτοι μήνες λοιπόν ήταν δύσκολοι, δεν ήταν εύκολο να συναρμολογήσουμε τα κομμάτια του παζλ, αλλά όπως είπε και ο Πιέρ, στο τέλος του πρώτου έτους ε, μπορούμε με ικανοποίηση να πούμε πώς καταφέραμε να δημιουργήσουμε δομές και διαδικασίες ε, ενός ε, υγιούς οργανισμού. Προσλάβαμε 150 άτομα από 6.000 αιτήσει. Συμφωνώ με τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Σεύκοβιτς πως έχουμε καλή σχέση εργασίας με την Κομισιόν και αυτό φαίνεται από την ε, συνεργασία στην πολιτική, είτε μιλάμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είτε για την πολιτική γειτονία, αλλά και σε πιο καθημερινά πράγματα. Έχουμε νέες δομές για το κοινό μας προσωπικό στις αντιπροσωπείες και μοιραία υπήρχαν κάποιες εντάσεις και γραφειοκρατικές διαφωνίες, αλλά Νομίζω πως καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτή τη φάση και τώρα έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τους συναδέλφους ε, της Κομισιόν και στις Βρυξέλλες και στις αντιπροσωπείες. Βεβαίως ε, πρέπει να αναλάβουμε και το έργο της ε, κυλιόμενης Προεδρίας στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στα οποία τώρα προεδρεύει η υπηρεσία και να έχουμε σχέσεις με την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και βεβαίως στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και μέσω της ε, κάθε άστων που αποδίδει μεγάλη σημασία σε αυτό, αλλά βεβαίως και η επικεφαλής αντιπροσωπιών και τα λοιπά είναι στη διάθεση των βουλευτών και προσπαθήσαμε να δούμε με λιγότερη επιτυχία το ομολογώ το ζήτημα των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων Επιπλέον ε, έπρεπε να αποκτήσουμε σχέσεις με τον Όλαφ, ε, το Μεσολαβητή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος ο κ. Σεύκοβιτς έπρεπε να στηρίξουμε και τους Προέδρους Μπαρόσο και Φαν Ρόμποϊ υπό την ιδιότητά τους ως εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συνόδου της Μέσης Ανατολής. Όλα αυτά ήταν μια πρόκληση λοιπόν και σίγουρος πως οι διαδικασίες που έχουμε δεν είναι τέλειες αλλά τώρα έχουμε ένα μοντέλο εργασία το οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε ελπίζω στο μέλλον. Βεβαίω έπρεπε και να φροντίσουμε το δίκτυο των αντιπροσωπιών. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα διπλωματικά δίκτυα στον κόσμο. Ε, έκτο νομίζω μετά τις ΗΠΑ, ε, Κίνα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία. Μεγάλο πλεονέκτημα για την υπηρεσία ναι, έχουν βεβαίως και μεγάλη συνεισφορά από τους συναδέλφους της Κομισιόν. Εξακολουθούμε να θεωρούμε πως ε, τα οικονομικά των αντιπροσωπιών δεν είναι τέλεια, δεν συμφωνούμε πλήρως με την ε, Κομισιόν και με βουλευτές βεβαίως. Ξέρω πως δεν έχουμε την ίδια άποψη, οπότε θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά για να ενσωματώσουμε πλήρως τις αντιπροσωπίες στο έργο της υπηρεσίας ε, έτσι ώστε να μην εφαρμόζουν μόνο οδηγίες από τις Βρυξέλλες αλλά να διαμορφώνουν την πολιτική. Ένα, μια αλλαγή δηλαδή στο πώς ε, στο σκεπτικό των αντιπροσώπιων και η εμπειρία που ανέφερε ο Πιέρ ε, με την συνεργασία επιτόπου με τις πρεσβείες των κρατών μελών είναι πάρα πολύ θετική και νομίζω πως υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για συνέργεια και εξοικονόμηση πόρων ε, π.χ. το να μοιραστούμε χώρους, ε, το να υπάρχουν ε, διπλωμάτες με ένα λάπτοπ στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ωφελήσουν και εμάς και τις εθνικές διπλωματικές αρχές. Επίσης έχουμε ένα νέο κτίριο και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για αυτό. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι μιας νέας διοικητικής νοοτροπίας και θα υπάρχει έτσι και μια αίσθηση ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από πολλές υπηρεσίες ε, ότι ανήκουν σε μια υπηρεσία. Θεωρώ λοιπόν πως έχουμε επιτύχει πολλά μέσα σε ένα χρόνο. Ε, πρόκειται για κάτι το μέσο μακροπρόθεσμο. Θεωρώ πως θα χρειαστούμε ακόμα 3-4 χρόνια για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και σε τελική ανάλυση αυτό είναι το υλικό, αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί ότι θα δημιουργήσει κάθε άστον ε, ως πρώτη ε, είπατε Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ικανή σύγχρονη διοίκηση. Βεβαίω το λογισμικό, αν θέλετε, τελικά είναι η διάθεση να χαραχθεί πολιτική. Και εδώ πέρα λοιπόν έχουμε την καινοτομία όσον αφορά το υλικό με την νέα αυτή υπηρεσία αλλά δεν έχει αλλάξει κατά πολύ το λογισμικό μέσω της Λισαβόνας, ε, καθώς μιλάμε ακόμα για ομοφωνία στον τομέα της ΚΕΠΑ και θα προσπαθήσουμε εδώ πέρα να επιδείξουμε ένα, έναν ηγετικό ρόλο, αλλά βέβαια αυτό εξαρτάται και από το πόσο θέλουν να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη. Να μιλάνε δηλαδή με μία φωνή σε ζητήματα διεθνή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, David. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και τους αντιπρόεδρους της Επιτροπής για την πρόσκληση. Όπως θα ξέρετε, ε, το ελεκτικό συνέδριο ε, ε, παρά κάποιες μικρές επικρίσεις κατέληξε σε πολύ θετικά συμπεράσματα για, τις, για τον ρυθμό ε, της παροχής βοήθειας και της διαδικασίας δημοσιονομική διαχείρισης. Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτές τις βελτιώσεις ε, και να μην τις ε, υπονομεύσουμε σε καμία περίπτωση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία. Καταρχήν, οι ρυθμίσεις είναι αρκετά περίπλοκες και μετά θα αναφέρω και μερικά πρακτικά παραδείγματα για τα έμπρακτα αποτελέσματα του νέου θεσμικού πλαισίου καταλήγοντας σε μερικές πρόσφατες εξελίξεις, αν προλάβω. Καταρχήν λίγα λόγια για την περιπλοκότητα των ρυθμίσεων. Είναι σαφές ότι η σύσταση της ΑΕΔ έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, ε, στο τοπίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλαξε ξεκέλευθε και την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Οι αναπτυξιακές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, συμπεριλήφθηκαν στην ΤΕΦΚΟ που είναι ο βασικός εταίρος της ΑΕΕΘ πια και ταυτόχρονα με τη σύσταση της ΑΕΕΘ τα μέσα και μηχανισμοί εξωτερικής πολιτικής ε, επίσης ιδρύθηκαν και η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει την υπατή εκπρόσωπο. Πέραν της ΔΕΦΚΟ, η FPI ε, ασχολείται με την διεύρυνση, το ΕΚΟ και το εμπόριο. Αυτό είναι το πλαίσιο δηλαδή που σημαίνει ότι είναι δυνατόν οι επικεφαλής αντιπροσωπιών να έχουν επαφές ταυτόχρονα με τέσσερις διαφορετικές υπηρεσίες ε, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν δούμε την, καταμερι... την κατανομή αρμοδιότητα μεταξύ της ΕΙΕΔ και της ΔΕΦΚΟ για βασικά θέματα όπως είναι ο προγραμματισμός, βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποιες ασάφειες σε αυτόν τον καταμερισμό των ε, ευθυνών και των αρμοδιοτήτων. Στις 13 Ιανουαρίου του 2012 είχαμε νέες ρυθμίσεις για την διευκρίνηση της κατανομής αυτών των ευθυνών και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι ότου αξιολογήσουμε αυτές τις νέες ρυθμίσεις. Το νέο καθεστώς των αντιπροσωπιών ως ε, Ιωνί πρεσβείες και των ε, επικεφαλής αντιπροσωπιών ως πρεσβευτών επίσης ε, δίνει έμφαση στον πολιτικό ρόλο. Κάτι που αναγνωρίζεται γενικώ, αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνει τους επικεφαλής αντιπροσωπιών γιατί θα πρέπει ταυτόχρονα να επιτελούν δύο διαφορετικά καθήκοντα και είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέρχονται σε αυτό το διπλό ρόλο, τον πολιτικό και τον διοικητικό. Τώρα, ένα άλλο σημείο είναι σε ποιο βαθμό υπάρχει ε, αλλαγή των ε, η μετάβαση από τις πολιτικές ιδιότητες στις αναπτυξιακές και πώς ε, ο ίδιος υπάλληλο μπορεί να περνάει τη μία ιδιότητα στην άλλη, ιδιαίτερα σε εποχή που το προσωπικό είναι, το προσωπικό είναι πολύ λίγο μειωμένο και ταυτόχρονα εφαρμόζονται σημαντικές λειτουργίες και χρονοβόρες βέβαια, όπως ε, είναι ε, η ε, αξιωματούχοι και για, και για την ΕΕ και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα πρακτικά αποτελέσματα του νέου θεσμικού πλαισίου. Βέβαια δεν έχει ήδη ακόμη έλεγχος για το θέμα αυτό, αλλά έχουμε εξετάσει κάποια έγγραφα και μάλιστα την αντιπροσωπείες, συζητήσαμε με τους υπαλλήλους εκεί και αυτό που είδαμε στην πράξη είναι μία δυσφορία σε αντιπροσωπείες ως προς το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο. Και θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα έγγραφα. Μία απάντηση του Διευθυντού του Νοεμβρίου, δεν σας πω πότε ακριβώς, Ε, σε ό,τι αφορά δύο, εξωτερι... δύο εκθέσεις εξωτερικής, ε, διαχείρισης εξωτερικής ε, βοήθειας και λέει ότι σε ό,τι αφορά τη χρήση του προσωπικού λυπούμαστε γιατί δεν μπορούσαμε να οριστικοποιήσουμε τις ρυθμίσεις εργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΙΕΔ. Συνεχίζει η απάντηση ότι θα πρέπει το οι υπάλληλοι να επικεντρώνονται στις ε, συγκεκριμένες ε, ευθύνες τους άσχετα με το αίτημα για περισσότερη ελαστικότητα. Ένα άλλο παράδειγμα, σε έκθεση διαχείρισης ε, στα μέσα του προηγούμενου έτους αναφέρεται ότι η σύσταση της ΕΙΕΔ ως ξεχωριστής οντότητας δημιουργεί ένα κατακαιρματισμό στη διαχείριση των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό της ΕΕΔ θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει πλήρως στις επιχειρησιακές δραστηριότητες των αντιπροσωπιών και ε, οι ισχύοντες κανόνες είναι αναποτελεσματικοί για τις μικρές αντιπροσωπείες. Και τέλος ένα σύντομο τρίτο παράδειγμα, όπου αναφέρεται ότι η σύσταση της ΑΕΔ με ε, στελέχωση της, ε, των αντιπροσωπιών από την ΑΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σοβαρές συνέπειες στην εφαρμογή του των αναπτυξιακών προγραμμάτων του προγραμμάτων του Αναπτυξιακού Ταμείου. Επίσης αναφέρεται στη συνέχεια ότι για να αποφύγουμε εμπλοκή της αναπτυξιακής βοήθειας σε περιφερειακές ε, αντιπροσωπείες θα πρέπει να ελέγχονται τα έγγραφα αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς δυνατότητα να πραγματοποιούνται και επιτόπιοι έλεγχοι της κατάστασης. Αυτά είναι αποσπάσματα από εκθέσεις. Και παρόλο που αυτά αναφέρθηκαν στις 15 Μαρτίου στο, ε, στο κεντρικό γραφείο, δεν δόθηκε μία απάντηση. Φαντάζομαι θα υπάρχουν εύλογοι λόγοι για την καθυστέρηση αυτή της χωρίς απάντησης, αλλά δείχνουν ε, τις δυσκολίες στην πράξη. Έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, γι' αυτό δεν θα σας αναφέρω τις πρόσφατες εξελίξεις. Τους ή ε, έχω γραπτός και την ομιλία μου, θα μπορούσα καλύτερα να σας ε, την ε, δώσω. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Και... Κύριε σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση σε αυτή την ακρόαση. Θα κάνω μία σύντομη εισαγωγή με βάση μια έρευνα που είχα κάνει για τις αναδυόμενες χώρες και βασιζόμενος σε επαφές μου με συναδέλφους στην Αφρική και την Ασία. Ο τίτλος Έχω τέσσερις ε, διαφάνειες, τόσο ή είναι μικρές, δεν θα μπορέσετε να τις δείτε. Ο τίτλος είναι Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική Αναζήτηση Σημασίας. Αυτή για μένα είναι η πρόκληση. Τι εννοώ με αυτό ως βασικό πρόβλημα. Στην ε, συζήτηση ε, ανέφεραν οι ομιλητές ε, την ανάγκη να έχουμε ξεκάθαρες στρατηγικές. Η βασική μου ανησυχία είναι πως ξεχνάμε και η Υπηρεσία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως η βασική πρόκληση είναι πως τα υπόλοιπα μέρη του πλανήτη δεν θεωρούν πλέον σημαντική την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε ε, οι εξελίξεις σε 5, 10, 20 χρόνια, η αμφισβήτηση της σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν έχει σημασία αν έχουμε καλή στρατηγική για την ε, προώθηση τη δημοκρατίας, αν δεν μας ακούνε στον υπόλοιπο πλανήτη, δεν μας θεωρούν σημαντικούς. Δεν θα έχει αντίκτυπο αυτή η στρατηγική. Υπάρχουν τρία πράγματα λοιπόν που θα ήθελα να αναφέρω. Πράγματα τα οποία ξέρουμε, αλλά έχουν εντύπωση πως δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα το τι σημαίνουν ε, ως προς τις συνέπειε τους. Δεν βλέπετε καλά εδώ πέρα την ε, διαφάνεια, αλλά είναι ένας παγκόσμιος χάρτης ε, κινέζικος. Με την Κίνα στο κέντρο, η Ευρώπη βλέπετε είναι στην άκρη ε, και με κέντρο τον ειρηνικό και της είπα βεβαίως. Οπότε στις επαφές μου με Αφρικανούς και Ασιάτες συναδέλφους είναι σαφές πως θεωρούν αυτές τις χώρες τις ανερχόμενες και την Κίνα ως πιο θεμητές, ε, νόμιμες, αξιόπιστες φιλοδοξίες τους ε, και αποτελεσματικές. Και εδώ πέρα είναι το πρόβλημα, γιατί δεν θεωρείται αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη διαφάνεια, θα τα βρείτε αυτά και στα χαρτιά που σας έδωσα, έχουμε νέους ε, σχηματισμούς και δίκτυα ισχύω. Ήψα, BRICS, APEC, η συνεργασία της Αγκάης και άλλα που δεν ξέρουμε ακόμα έχουν εντύπωση πως όλα αυτά δεν οδηγούν σε κάποιο σαφές ε, συμπέρασμα. Στις επαφές μου με τους Κινέζους και Ασιάτες συναδέλφους, τα δίκτυα αυτά οδηγούν σε αποτελέσματα στη χάραξη πολιτικής αυτών των χωρών. Και αυτή είναι η πρώτη μου συμβουλή στην υπηρεσία για το μέλλον και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μην εστιάζετε σε χώρες μόνο, αλλά φροντίστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις συζητήσεις σε όλα αυτά τα άτυπα δίκτυα γιατί αυτό το οποίο έμαθα από τις Ασιάτες συναδέλφους είναι πως είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από όσο νομίζουμε. Επόμενη πρόκληση, ο λαός. Ξέρουμε πως είναι σημαντικός, μας αρέσουν οι επαναστάσεις στις διάφορες χώρες. Το πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να δώσει μια απάντηση στις ανάγκες του λαού. Ανεργία, βασικές ανθρώπινες απαιτήσει. Βασικό πρόβλημα εδώ πέρα είναι πως οι άνθρωποι αυτοί, όχι μόνο στις αραβικές χώρες, αλλά και στην Αφρική, είναι πως θεωρούν την Κίνα ως πολύ πιο σημαντική και αποτελεσματική χώρα που μπορεί να τους βοηθήσει. Ο κόσμος στις χώρες της Βορειοαφρικής ε, θεωρεί τα Ισλαμικά κινήματα πολύ πιο αποτελεσματικά Ισλαμικά κινήματα τα οποία συχνά στηρίζονται οικονομικά από τη Σαουδική Αραβία και άλλες ε, χώρες ε, του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Πρέπει να δούμε μια συνολική προσέγγιση. Δεν πρέπει να ξεκινάμε μόνο από τα μέσα τα οποία έχουμε εδώ πέρα στην Ευρώπη αυτά τα οποία ανέπτυξε η υπηρεσία εξωτερική δράση τα τελευταία δύο χρόνια και ξέρω βεβαίω πω αυτό είναι δύσκολο και έχει υπάρξει μια θετική διαδικασία, πρέπει να ξεκινήσουμε από την προοπτική των α, χωρών της άλλη πλευράς. Τι περιμένουν, τι, πώς μπορεί να δείξει τη σημασία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα λοιπόν εντολή σημαντική για την υπηρεσία και τις αντιπροσωπείες είναι ακριβώς να καταγράψει όλα αυτά τα πράγματα, να δούμε για την κάθε χώρα και περιοχή το τι στόχους έχουν, τι θεωρούν αυτοί σημαντικό, όχι το τι θεωρούμε εμείς σημαντικό. Δεύτερον, τι πολιτικές μπορεί να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δείξει πως έχει σημασία, γιατί μόνο όταν δείξουμε πως έχουμε σημασία μπορούμε να μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία. Το ερώτημα είναι μετά από αυτή την καταγραφή χρειάζεται και ένας οδικός χάρτης με σαφείς ε, προτεραιότητες που θα είναι όρατες. Αυτό έμαθα από τους συναδελφούς στην Αφρική. Οι Κινέζοι έχουν απτά αποτελέσματα, το ίδιο πρέπει να κάνετε και τι σημαίνει αυτό για την υπηρεσία εξωτερική δράση. Η υπηρεσία χρειάζεται πολύ περισσότερου έμπειρογνώμονε ε, στον αραβικό κόσμο, Κίνα, Ασία κτλ. Ανθρώπου θα ξέρουν κινέζικα, αραβικά ειδικού όχι στις ε, ευρωαραβικές σχέσεις αλλά στον αραβικό κόσμο και ξέρουμε βεβαίω πως ο προπολογισμό ε, του προσωπικού δεν θα αυξηθεί αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να συνεργαστεί με ειδικού από Think Tank ε, η υπηρεσία και βεβαίως πρέπει να αλλάξει η πολιτική στελέχωσης και του προσωπικού. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε κινέζικα στο Πεκίνο εργάζεται αυτή τη στιγμή για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης στην Τινησία. Δεν είναι δυνατόν. Τέλος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να παίξει ένα ρόλο. Πρέπει να εξηγήσουμε στο κοινό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη τα συμφέροντα τρίτων χωρών και των λαών τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες προηγούνται. Ο κύριο Αλαφράγκα, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι άσχετα με τα προσωπικά ζητήματα που επηρέασαν ε, το έργο της ΥΠΑ της εκπροσώπου, καλό θα ήταν να, να κάνουμε μια ε, αντικειμενική αξιολόγηση της πραγματικότητας και να επικεντρωθούμε στα θεμελιώδη. Το βασικό είναι ότι με τη σύσταση της ΕΙΕΔ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση με πολύ πιο αποτελεσματικό, ε, προβεβλημένο και αξιόλογο τρόπο να επιτελεί το έργο της και θεωρούσαμε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα της εξωτερικής πολιτικής εκεί σε Ανατολή Ιράν, ε, παγωμένες συγκρούσεις, ε, αν νομίζαμε ότι θα ε, λυθούν διαμαγείας, ήταν προφανές πως δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον έχουμε μια πιο συνεκτική δράση τη εξωτερική μα πολιτική χάρη στην ΕΕ. Ούτε ήταν εύκολο κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να επιθυμίσω εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήσαμε ε, να ε, ε, εμπίπτει η ΕΙΕΔ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελικά δημιουργήθηκε μια υβριδική οντότητα με διακυβερνητικά χαρακτηριστικά και μετά από τις ε, αρχικές διακοιμάνσεις που είχαμε με την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοινική Συνέλευση του ΟΗΕ τα προβλήματα τελικά που καλύφθηκαν. Προβλήματα στο για τη θέση της Παλαιστίνης στην UNESCO και η παρουσία της Παλαιστίνης στην, στις διεθνείς οργανώσεις, όλα αυτά δείχνουν ότι η σύσταση και η περαιτέρω ε, διεξαγωγή των εργασιών της ΑΕΣ ό,τι αφορά θέματα προσωπικού, τελικά ήταν μια επιτυχημένη προσπάθεια. Και μπορούμε να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό. Παρόλο που είναι προφανές ότι πολλά θα πρέπει ακόμη να γίνουν. Έχω την αίσθηση, κύριε Πρόεδρε, ότι το παράδειγμα της Αραβικής Άνοιξης είναι ένα θετικό παράδειγμα. Και εκεί υπήρξαν κάποιες αρχικές αμφιταλαντεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας όταν εγκρίθηκε το ψήφισμα για την ε, αποκλειστική ζώνη πτήσεων στη Λιβύη. Αλλά νομίζω ότι γενικώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε μια καλή εικόνα για την ε, εφαρμογή της ενισχυμένης πολιτικής ΙΕΣΥΣ. Πιστεύω ότι η ΕΕΔ δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε μια προσπάθεια ε, διελκυστίδας μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να ε, αποτελέσει ένα όργανο προς εξυπηρέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του, της εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λόγους να είναι ικανοποιημένο από τις ε, δεσμεύσεις που ανέλαβε η πρόσωπο και νομίζω που τις έχει επιτελέσει με μια μικρή εξαίρεση. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα αποτελέσματα του Υπουργικού Συμβουλίου Εξωτερικών. Προηγουμένως είχαμε την υπατεκπρόσωπο, την ε, ε, Προεδρία και τον Επίτροπο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Ο κύριος Φίλερ Χόταν τώρα έρχεται που και που η Προεδρία, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται ε, συνέχεια ενημέρωση στο κατάλληλο επίπεδο. Είμαστε ικανοποιημένοι, ε, αλλά πολλά ακόμη θα πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνει ένα ποιοτικό άλμα, να βελτιωθεί ο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και να υποβληθούν προτάσει όχι μόνο αντιδραστικές αλλά και ε, πρωτοβουλίας. Να μην αντιδρούμε μόνο, να ε, προτείνουμε και όλα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κοινοποιήσουμε αυτές τις θετικές παρατηρήσεις προς την ε, είπατε εκπρόσωπο με φυσικά σκοπό να βελτιωθεί η λειτουργία της ΕΕΔ. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. I also, and my group also makes... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ και η ομάδα μου εκτιμούμε θετικά το έργο σε αυτό το πρώτο χρόνο ε, εγκαθίδρυσης της ΕΕΔ και φυσικά με επικοδομητικό πνεύμα τονίζουμε τα στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση, πράγμα το οποίο είναι φυσιολογικό, διότι όπως ε, ήδη τονίστηκε, προφανώς ε, η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε ενώ ταυτόχρονα ξέσπαγαν ένα σωρό κρίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και άρα ήταν φυσιολογικό να είναι δύσκολη αρχή. Με αυτή την ε, επικοδομητική λοιπόν ε, προσέγγιση θα αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία μέσω των το εκπροσώπου μας που ήταν ήδη εκεί από την αρχή με τον Ρομπέρτο Γουαλτιέρη που δυστυχώς σήμερα δεν είναι εδώ Θα τον αφήσω εκείνο να κάνει την πολλή δουλειά. Πάντως θα πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι με επικοδομητικό πνεύμα τονίζουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που βλέπουμε και που μπορούν να διορθωθούν και πρέπει να διορθωθούν, διότι ε, θέλουμε να δώσουμε αυτό το ευρύ πνεύμα αρμοδιοτήτων στην ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αλλά και να έχουμε και αυτή την στρατηγική προσέγγιση που ανέφερε ο πρέσβης Βήμου, ότι δηλαδή το στρατηγικό όραμα που τονίζει προτεραιότητες δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, μπορούμε να κάνουμε πολλά όμως και πρέπει να έχουμε προτεραιότητες στρατηγικές. Πιστεύω λοιπόν ότι τα προβλήματα κυρίως έχουν να κάνουν με τις σχέσεις με την Κομισιόν Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα που θα μπορούσα να σας αναφέρω εδώ, αλλά δεν χρειάζεται να τα αναφέρω όμως. Απλά να τονίσω την έλλειψη εφαρμογής από πλευρά της Κομισιόν των όσων συμφωνήθηκα στη Μαδρίτη για τη μεταφορά στην υπηρεσία της μονάδας της Επιτροπής που ασχολείται με το μέσο σταθερότητα. Ένα άλλο στοιχείο είναι η αποτελεσματικότητα της αλυσίδας της ιεραρχίας Υπάρχει ένα πρόβλημα ανάμεσα στον Γενικό τον εκτελεστικό γραμματέα και τον διοικητικό διευθυντή. Δεν είναι ακριβώς η συνεργασία που θα έπρεπε να υπάρχει. Και αυτό επηρεάζει το συντονισμό, τη συνοχή και τη συνέπεια όσον αφορά την αλληλουχία των διαφόρων βαθμίδων. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μια δημοσιονομική κρίση όπου τα κράτη-μέλη μας θα μπορούσαν να πούν ένα σωρό πράγματα αλλά δεν έχουμε κάποιον ε, στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ και δεν έχουμε ωστόσο κάποιον, κάποια ηγετική φυσιογνωμία στο πλαίσιο της ΕΙΕΔ ε, που θα υποστηρίζαμε αν πίεζε τα κράτη-μέλη πως ε, κάτι συγκεκριμένο χρειάζεται. Γιατί αυτή είναι και η λειτουργία, να μην ευνοεί τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου κράτους μέλους, αλλά να προωθεί τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και όσον αφορά τις εξωτερικές δράσεις, όπως τόνισε δικαίως ο κύριος Κέικελερ. Επίσης υπάρχει το θέμα της ισορροπίας ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς υπάλληλους και τους κρατικούς υπάλληλους δεν θέλω αυτό να μετατραπεί σε έναν ανταγωνισμό. Ζητήσαμε μελέτες για την γεωγραφική ισορροπία και την ισορροπία των φύλων, αλλά φυσικά η αξιοκρατία θα πρέπει να επικρατήσει, αλλά και τα προσόντα και κυρίως ε, τα γλωσσικά προσόντα των υποψηφίων. Και φυσικά έχουμε και το θέμα της δημοκρατικής, ε, του δημοκρατικού ελέγχου, της λογοδοσίας. Έχουν γίνει πολλά, το εκτιμούμε πολύ αυτό την ε, επαφή δηλαδή με την υπηρεσία, αλλά και πάλι αυτό είναι ένας τομέας όπου θα έπρεπε να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις για ένα στρατηγικό διαλόγη Βέβαια ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα εξετάσουμε αυτά περαιτέρω. Ευχαριστώ. Uh, Mr. President, your colleagues, uh, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω το πόσο εκτιμούμε την ακρόαση αυτή. Δεύτερον, θα ήθελα να μοιραστώ το χρόνο ομιλίας με τους άλλους συναδέλφους από την αντιπροσωπεία που ζήτησαν να μιλήσουν. Θα είμαι λοιπόν σύντομη. Είμαι σύντομη, θα πω λίγα πράγματα. Πρώτα απ' όλα όταν η Βαρόνια στον ήρθε εδώ πέρα μας υποσχέθηκε πως θα έφτιαχνε μια υπηρεσία πριν το τέλος του έτους. Τότε πολλοί αμφέβαλαν για το αν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Τα κατάφερε όμως. Μέχρι το τέλος του έτους ή τέλος πάντων τις πρώτες μέρες του επομένου έτους η υπηρεσία είχε στηθεί, εντάξει μπορεί να μην λειτουργούσε αλλά δούλευαν οι άνθρωποι εν πάση περιπτώσει και αυτό από μόνο του κάτι είναι. Δεύτερον, το ότι λειτουργήσε στα διάφορα γεγονότα που όλοι ε, γνωρίσαμε ε, είναι επίσης κάτι το εξαιρετικό. Τρίτον, έχασα το, τον ήρμό μου. Ναι, Κάτι το φανταστικό λοιπόν. Τρίτον, ναι. Much we would like, uh, the service to prioritize. Όσο και αν θέλουμε να δίνει προτεραιότητες η υπηρεσία σε κάποιες περιοχές, παρόλα αυτά θα θέλαμε πάντα να συνειδητοποιούμε πως ο κόσμος έχει τον τρόπο του να μπαίνει ε, στο σκηνικό και θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Και βεβαίως το Κοινοβούλιο αναμένει από την ε, είπατε εκπρόσωπο να μιλάει και να μιλήσει σύντομα βεβαίως, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εύκολα συμβατό. πρώτη μας προτεραιότητα είναι η γειτονιά μας η αυλή μας, αν θέλετε. Μπροστά ή πίσω αυλή δεν έχει σημασία. Και η βασική μας ευθύνη. Τέλος, μου επιτρέπετε να πω κάτι σε έναν από τους προλαλήσαντες. Εγώ προσωπικά θα σοκαριζόμουν εάν η Βαρώνη ε, στο προσεχές μέλλον Ε, μπορούσε να κάνει σε έναν από τους ε, κύριου εκφραστές εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο έκαναν οι κινέζικε αρχές στον Μπότσι Λάι. Yes, thank you, Chair. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη δική μου ομάδα θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι στην αρχή όλοι γνωρίζαμε πως η ΑΕΔ θα είναι μια δύσκολη επιχείρηση για όποιον και την αναλάβει και παρά τις αδυναμίες ε, και τα εμπόδια που προέκυψαν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, γιατί δεν είναι κανονικό Υπουργείο, δεν είναι κανονικό Γραφείο Εξωτερικών Σχέσεων, δεν είναι πλήρες Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά είναι αυτό που έχουμε. Είναι μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και παρά τα εμπόδια και τις αδυναμίες που υπάρχουν, πιστεύω ότι παρόλα αυτά η ΕΕΔ έχει επιτελέσει αξιοθαύμαστο έργο. Είναι η έκτη σε μέγεθος υπηρεσία εξωτερικής δράσης στον κόσμο, όπως είπατε κι εσείς. Και η αποδοχή των αντιπροσωπιών αυτών από τα κράτη-μέλη και η υποδοχή των αντιπροσωπιών στις τρίτες χώρες είναι σχετικά θερμή. Και μάλιστα οι αντιπροσωπείς αυτές εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μεμονωμένα κράτη-μέλη. Όλα αυτά είναι επιτέγματα. Έχουμε τώρα τους τρεις άξονες, Κομισιόν, ε, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και κράτη-μέλη. Ούτε ε, και η συνεννόηση μεταξύ τους είναι εύκολη και αυτό και είναι λογικό να υπάρχουν δυσκολίες και στο μέλλον. Τώρα, συνεργασία μεταξύ αντιπροσωπιών και πρεσβειών των χωρών μελών. Υπάρχει ένα νέο σύστημα, το άσυντα, δεν κάνω με ε, κατάρτιση κοινών εκθέσεων από τις πρεσβείες των κρατών μελών. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας ε, από μια τέτοια πρόταση. Επίσης θα ήθελα η ΕΕΔ να πρωτοστατήσει στην διαμόρφωση της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ε, εξωτερικών υποθέσεων και στις διάφορες αντιπροσωπείες να είναι πρωτοπόρα στην, στον καθορισμό του πολιτικού προγράμματος από κοινού με τα κράτη-μέλη και μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα τα θέματα τα κράτη-μέλη όπως σε περιπτώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάντως συμφωνούμε, πιστεύω ότι όταν συμφωνεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα πρέπει οι επικεφαλείς των αντιπροσωπιών ε, να θεωρούν ότι έχουν το πράσινο φως ε, και να μπορούν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Θέλουμε τέτοια πρωτοκαθεδρία και πρωτοπορία από τις ε, αντιπροσωπείες. Επίσης, μπορεί να βελτιωθεί η παρουσία των γυναικών σε υψηλό επίπεδο. Έγιναν κάποιε προσπάθειε και βελτιώσει, αλλά δεν αρκεί. Περισσότερη παρουσία των γυναικών, ιδιαίτερα στα υψηλά κλιμάκια. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κρίσεων, είπατε κύριε Βημό ότι βάλαμε το πλοίο στη θάλασσα και ήδη έχει ξεκινήσει. Το θέμα είναι ε, πότε θα μπει στο λιμάνι και σε ποια κατάσταση θα μπει στο λιμάνι. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Θα υιοθετηθεί μια πιο σφαιρική προσέγγιση ό,τι αφορά την πρόληψη, διαχείριση των κρίσεων και την αποκατάσταση της ειρήνης. Γιατί ε, θα πρέπει να έχουμε και μη στρατιωτικό σημαντικό παράγοντα, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότερες ε, ε, δυνατότητες προγραμματισμού στα πλαίσια της ΚΕΠΑ έχουν και το προσωπικό έχει στρατιωτική σταδιοδρομία, παρόλο που οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μη στρατιωτικού χαρακτήρα. Αναφερθήκατε σχέσεις ΕΙΕΔ και ΝΤΕΦΚΟ. Εκεί υπάρχουν κάποιες ασάφειες για τις αρμοδιότητες του καθενός. Επίσης έχουμε τη μη κυβερνητική οργάνωση για την ανάπτυξη, την Concord. Εκεί υπάρχει εντύπωση ότι η ΕΙΕΔ δεν ενδιαφέρεται και πολύ για αναπτυξιακά θέματα. Πώς πιστεύετε εσείς ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον. Well, um, one year on, yes. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, ένα χρόνο μετά. Η ΕΕ, μάλλον η ομάδα μας βασικά συμφωνεί με την ΕΕ. Έχουμε οικοδομητικό στόχο. Νομίζω πως ε, ε, πρόβλημα ήταν η Λιβύη, αλλά τα ε, καλύτερα τα πήγαμε το Ιράν. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα πρέπει να μας εντυπωσιάζει δεδομένης της οικονομικής κρίσης που περνάει η Ευρώπη για τη διάσωση του ευρώ, πράγμα που έχει αποσπάσει την προσοχή των ηγετών των κρατών μελών από τα διάφορα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Γενικά ήταν δύσκολη χρονιά και δεν είναι πολύ εντυπωσιακό που η ΕΕΔ κατά κάποιο τρόπο μπήκε σε δεύτερο πλάνο. Ωστόσο, είναι, πολύ, ε, είναι εξαιρετική η δουλειά του, David, ε, του Pierre και του David O'Sullivan. Έφτιαξαν μια ολόκληρη υπηρεσία που ενώ διαδέχθηκαν ένα δίκτυο της Ένωσης ε, που βασικά ήταν αφιερωμένο σε εμπορικά θέματα και θέματα ανάπτυξης και όχι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Θα πρέπει ωστόσο να επανεξετάσουμε τα διάφορα θέματα. Ξέρω ότι υπάρχει ας πούμε μια ε, μεγάλη αντιπροσωπεία στα υπέροχα και εξωτικά Μπαρμπάδος, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχα σοβαρή αντιπροσωπεία στον Παναμά που αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία. Θα πρέπει κάποια τέτοια πράγματα θα διορθωθούν. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει περιορισμός από πλευρά των κρατών μελών στις διμερείς τους αποστολές, ιδιαίτερα για τις μικρές χώρες. Ε, έτσι θα ποιωθεί το κόστος και έτσι θα μπορέσουμε να πλασάρουμε και καλύτερα την ιδέα της ΕΙΕΔ ως πιο αποτελεσματικής και οικονομικής. Ευχάριστη έκπληξη ήταν ότι δεν υπάρχει δυσαρέσκεια που ο Ευρωπαίος ε, πρέσβης ε, καταλαμβάνει την ε, μόνιμη θέση, μια μόνιμη θέση στις διάφορες συνεδριάζεις, αντί να έχουμε τον εκπρόσωπο της εκπεριοτροπής προεδρίας εκεί. οι υποψήφοι και οι οποίοι ε, εξετάστηκαν και προσλήφθηκαν ε, ε, στις θέσεις πρέσβεων ήταν εξαιρετικής ποιότητας και φυσικά υπήρξε μέγας σεβασμός και διευκόλυνση για τους ευρωβουλευτές ήρθατε σε επαφή μαζί μας σε ένα σωρό θέματα, πράγμα που δεν είχε παλιότερα εφαρμοστεί και έχουμε και γι' αυτό πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι πιο αναμεκτικό όταν ταξιδεύουμε σε τρίτε χώρε. Κάποιε φορέ οι Ευρωπαίοι πρέσβει και αντιπροσωπείε υποστηρίζουν, ενώ κάποιε φορέ λείπουν παντελώ. Απουσιάζουν. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Εγώ νομίζω ότι θέλουμε να υπάρχει με, να απαιτούμε μάλλον ε, ουδετερότητα δημοσιονομική, αλλά μετά από μια χρονιά θα πρέπει να σα πω ότι ήταν ευχάριστη έκπληξή μου για διάφορου τομεί και αντίθετα από την κυρία Λουνατσέκ, εγώ καλωσορίζω την, τον ρόλο ε, των ε, ε, αντίδρασης που έχει κρατήσει πολλές φορές η πατή εκπρόσωπος. Προτείνω να ακούσουμε κάποιες πρώτε και μετά να ε, περάσουμε σε έναν άλλο γύρο ερωτήσεων. Η Κομισιόν λοιπόν πρώτα. Ε, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ πως ο πρώτος γύρος ε, παρεμβάσεων επιβεβαίωσε πως Έχουμε επιτύχει σημαντική πρόοδο και συμφωνώ πλήρως με τον David πως η αρχή δεν ήταν εύκολη ούτε για την υπηρεσία μας ούτε για την Κομισιόν γιατί και εμείς έπρεπε βεβαίω να κάνουμε σημαντική αναδιάρθρωση αλλά τώρα θεωρώ πως είμαστε σε μια φάση όπου βλέπουμε πως η υπηρεσία αυτή ε, και η Κομισιόν ενισχύουν αλλήλους. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε και θα ήθελα λίγο να το αναφέρω, ένα σημαντικό τμήμα της συνεργασίας μας, η εξωτερική διάσταση σε πολύ σημαντικές εσωτερικές πολιτικές της Ένωσης. Βλέπουμε πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον των εταίρων μας για τις πολιτικές ενέργειας, περιβάλλοντος, ε, εμπορίου, καινοτομίας, έρευνας, γιατί μας θεωρούν ε, σημαντικούς παγκοσμίως και υπάρχει ε, ήδη επιθυμία από τους εταίρους μας να συνεργαστούμε. Οπότε έχω κάποιο πρόβλημα να δεχτώ πλήρως την ανάλυση του κυρίου καθηγητή. Γιατί αντιλαμβάνομαι πως το βλέπει από μια ακαδημαϊκή σκοπιά, αλλά από μια πρακτική σκοπιά δεν θεωρώ πως έχουμε πρόβλημα σημασίας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για τις ανερχόμενες οικονομίες, αλλά ξεχνάμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμη μια μισή φορά μεγαλύτερη από όλες τις BRICS μαζί. Και όταν μιλάμε για εμπορικές σχέσεις, είμαστε το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ του πλανήτη. Και μεγαλύτερος εξαγωγέας, ε, με τις περισσότερες εφευρέσεις και πιο ελκυστική για τις ξένες επενδύσεις. Και δείχνει αυτό το πόσο ο ρόλος μας έχει βελτιωθεί και στις ομάδες G8, G20, σε όλες τις εμπορικές συνομιλίες, παρά το ότι βλέπουμε πόσο πολυμερείς γύρω στις Ντόχα δεν πηγαίνει με το ρυθμό που θα θέλαμε, αλλά βλέπουμε μια ξεκάθαρη απέτηση από τους εταίρους μας να έχουμε συγκεκριμένες διμερείς συνομιλίες και αντιμετωπίζουμε ε, ακριβώ αυτά τα αιτήματα και δεν έχουμε αρκετό προσωπικό για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τι διαπραγματεύσει. Οπότε όταν μιλάμε για όλα αυτά τα ζητήματα, για το τι κάνει η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αφρική, πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτά τα οποία κάνουμε εκεί πέρα. Ότι κάνουμε βασίζεται σε σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπέρ της ε, αηφόρου ανάπτυξης, ε, της ε, χρηστής διοίκησης και βεβαίως της υπευθυνότητας όσον αφορά τον προπολογισμό, γιατί είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Οπότε πράγματι υπάρχουν όροι σε αυτά τα οποία κάνουμε, αλλά πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί αυτή η όρη είναι η αξία μας, μας και πρέπει να το δούμε και από αυτή τη σκοπιά, γιατί εντυπωσιάστηκα από τα σηματάκια διαφόρων ομάδων εδώ πέρα που παρουσιάσατε στην ε, διαφάνεια αυτή, αλλά αν δείτε, αν πάτε σε μια σύνοδο, το πώς είμαστε εμείς προετοιμασμένοι και το πώς είναι αυτές οι ομάδες, ε, μη συγχαίουμε τώρα ομάδες που συναντιόνται μια φορά το χρόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και καμιά φορά έτσι υποδημούμε και τον εαυτό μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω σε μερικές ερωτήσεις και τις πιο δύσκολες θα τις αφήσω για τον Ντέιβιτ. Τώρα, για τη σχέση με την Επιτροπή, συμφωνώ απόλυτα με τον Επίτροπο. Όλοι συμφωνούμε ότι Υπάρχουν όλο και περισσότερες αναδυόμενες οικονομίες και χώρες. Φυσικά είναι γνωστό γιατί ο κόσμος αλλάζει, η διεθνής κοινότητα αλλάζει και δεν είναι κακό αυτό γιατί ε, έχουμε νέες ε, χώρες πολύ ανταγωνιστικές που διεκδικούν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο τώρα για τη σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τα οικονομικά στοιχεία που μας δίνουν ότι έχει ειδικό βάρος και μεγάλη σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παγκόσμιο προσκήνιο. Και αν περάσει κανείς από το γραφείο μου θα δει πόσες επισκέψεις έχουμε καθημερινά. Βέβαια πολλές φορές μας ζητούν απλώς χρήματα, αλλά πολλές φορές μας ζητούν και πολιτική καθοδήγηση. Αν δείτε τι έγινε με την Αραβική Άνοιξη, θα, θα διαπιστώσει τι ακριβώς ρόλο καλείται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι προστιθέμενη αξία έχει η πανευρωπαϊκή δράση σχέση με την εθνική. Αφήνουμε να την πόρτα με την Αραβική Άνοιξη και στην Αφρικανική Ένωση, παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και καλά, παρά τις πολλές επιφυλάξεις των χωρών της περιοχής. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να γίνει μια γέφυρα που ε, διατήρησε τις επαφές μεταξύ των χωρών και μεταξύ των ομάδων χωρών στην Αφρική και αυτό ήταν πολύ χρήσιμο δεν είναι μόνο θέμα σημασίας και σπουδαιότητας. Είναι το πώς θα διαμορφώσουμε το νέο ρόλο, ε, τη νέα θέση και τη νέα αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το νέο κόσμο, τον συνεχώς μεταβαλλόμενο. Και αυτή είναι σημαντική πρόκληση, μίζων. Αλλά είναι διαφορετικό αυτό από το κατά πόσο θα πρέπει να προβληματιζόμαστε αν έχουμε κάποια σπουδαιότητα ή όχι. Η κυρία Γκόμες μίλησε για την κοινή ευθύνη και συμφωνώ μαζί της ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, αλλά υπάρχουν περιπλοκές όχι μόνο των εξαιτία των κρατών μελών, γιατί και τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν θα πρέπει να συμβάλλουν και να μοιράζονται. Ε, αλλά διανύουμε και μια σημαντική χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που μας περιορίζει μεν, αλλά και μας βοηθάει να αντιληφθούμε ότι τώρα, θα πρέπει να συνενώσουμε ε, τους σπόρους μας. Και όταν μιλούμε για συμβολή και μοιρασιά. Εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τι επιχειρήσει και τον ιδιωτικό κλάδο. Και αυτό είναι πιο περίπλοκο γιατί ο ιδιωτικό κλάδο, οι ιδιωτικέ επιχειρήσει χρειάζονται εγγυήσει, θέλουν να αισθάνονται ε, εμπιστοσύνη και σιγουριά για να εμπλακούν και αυτή η διαδικασία είναι πιο χρονοβόρα. Πάντως η κατεύθυνσή μας, η πορεία μας είναι σωστή. Και αν δείτε που πάμε αυτή τη συμβολή και τη μοιρασιά, το pooling and sharing, βλέπουμε ότι προχωρούμε πολύ καλά και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε γελοί ή ασήμαντοι στα προγράμματα που εγκρίνουμε. Και θα φανεί και στο στην επόμενη διάσκεψη κορυφή του ΝΑΤΟ στο Σικάγο. Και η κυρία Λούνατσεκ μας ρώτησε για τη διαχείριση των κρίσεων και με ρώτησε και πού βρίσκεται το πλοίο. Το πλοίο βρίσκεται στη θάλασσα. χρειάστηκε πολύ καιρό για να επιβιβάσουμε όλο το πλήρωμα και τους επιβάτες, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε επιτυχημένη φάση και όταν οργανώνουμε διάφορες πλατφόρμες Συρία και αλλού, όλοι συμμετέχουν, όχι μόνο η ΑΕΔ, e αλλά και οι συνάδελφοι από την ΕΚΟ, την Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και από άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμη και από το Συμβούλιο. Ε, όλοι δίνουν το παρόν, γιατί σε τέτοιες πλατφόρμες επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε και ε, επιδεικνύουμε όλο και πιο θετικό και συνεργάσιμο πνεύμα. Και αυτό είναι προς όφελος όλων μας. Και χρειάστηκε χρόνος για κάτι τέτοιο. Γιατί έχει αλλάξει το μεταξύ νοοτροπία. Αρχικά δεν ε, είχαμε αυτή την νοοτροπία τη σωστή ε, διαχείριση των κρίσεων και ως προς αυτό σημειώσαμε πρόοδο. Φυσικά πολλά ακόμη θα πρέπει να γίνουν και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το, τη μη στρατιωτική συνιστόσα της ε, ΚΕΠΑ. Πολύ σωστά το επισημάνατε και πολύ συχνά χρησιμοποιούμε στρατητικούς ε, γιατί εκεί υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη για προγραμματισμό τέτοιου είδους ε, επιχειρήσεων. Αλλά το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και που επισημαίνει πολύ συχνά και είπατε εκπρόσωπος, είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι ότι ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να διεκπαιρεώσουμε τις διάφορες ε, επιχειρήσεις και ΚΕΠΑ στο Κωσυφοπέδιο, τη Γεωργία, το Αφγανιστάν ή αλλού. Ταυτόχρονα θέλουμε να ξεκινήσουμε και νέες επιχειρήσεις χωρίς ε, μερικές φορές ε, ε, να έχουμε αρκετούς πόρους και να μην δείχνουμε ότι μας λείπουν οι πόροι, γιατί θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι. Όταν συναντιόμαστε με τους συναδέλφους του ΝΑΤΟ και μιλούμε για το κοσυφοπαίδιο, το ότι δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε για τις αστυνομικές μονάδες, η εντύπωση που δίνουμε είναι ε, αρνητική, δημιουργείται μια ανησυχία για να μην πω τίποτα χειρότερο. Οπότε από αυτή την άποψη σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά θέματα, θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω τα λεγόμενα της είπα της εκπροσώπου στην ε, Επιτροπή Ανάπτυξης, που είπε ότι έχει επίγνωση του γεγονότος ότι είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει ταυτόχρονα σε όλες τις αποστολές της. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα ε, με τη διπλή ιδιότητα της είπα εκπροσώπου, αντιπροέδρου, προέδρου της, του, Υπουργείου Εξωτερικών, του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και με τόσες πολυάριθμες μετακινήσεις. Έχουμε τις εκπεριτροπής προεδρίες και τις εκπεριτροπής υπουργούς. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εφαρμόζεται όλο και περισσότερο Πάντως, μην ξεχνάτε ότι το 2011 η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος επισκέφθηκε πάνω από 36 χώρες, έκανε πάνω από 56 αποστολές και αυτή είναι η πραγματικότητα για την ΑΕΔ. Ο κύριος Αλαφράνκα υπογράμμισε κάποιες ε, ε, κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τις ε, τακτικές ενημερώσεις και του, του Υπουργικού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μπορεί να είναι πανταχού παρούσα η υπατή εκπρόσωπος. Προσπαθούμε ε, να ανταπεξέλθουμε στην υποχρέωση πολιτικής λογοδοσίας σε όλα τα συμβούλια αυτά και ευελπιστώ ότι θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες μας στην πορεία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, good for on minutes. Ευχαριστώ πολύ. Να ξέχασα να σας πω ότι θα πρέπει να μένετε στα πέντε λεπτά για τις απαντήσεις σας. Η Άννα Γκόμες είπε ότι δεν ήταν απόλυτα βέβαιη ότι ε, ο κύριος Βίμον, και εγώ θα συνεργαζόμασταν τόσο καλά, αλλά βλέπετε πόσο ωραία τα πάμε. Εκείνος απαντάει τις εύκολες ερωτήσεις και μου πετάει εμένα τις δύσκολες. Ε, καταρχήν να σας πω την αλήθεια πως ως υπηρεσία χρειάστηκε να αναλάβουμε πλήρη ευθύνη απέναντι στο ελεγκτικό συνέδριο και άλλα σώματα για τη δική μας διαχείριση. Δηλαδή όταν ήμασταν τμήμα της, ε, πράγμα το οποίο μάλλον όταν ήμασταν τμήμα της Γραμματείας του Συμβουλίου ή της ε, Κομισιόν δεν χρειαζόταν να το κάνουμε. Μάλιστα εγώ είχα μια πολύ καλή συζήτηση ε, με το ελεγκτικό συνέδριο ε, και νομίζω πως ε, τους έδειξα ότι θέλουμε να έχουμε μια σύγχρονη διαχείριση της υπηρεσίας μας και φυσικά θα διαβάσω την ομιλία σας στη γραπτή κύριε Πίνγκστεν γιατί στην αρχή υπήρξε, επικράτησε κάποια σύγχυση, δεν το αρνούμε. Υπήρχαν διάφοροι εξάλλου που οι υπάλληλοι της ΕΙΕΔ που δεξιά και αριστερά έλεγαν ότι δεν πάνε όλα ε, όπως πρέπει. Δεν λειτουργούν όλα τέλεια, ενώ νομίζω πως τώρα έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Έχουμε φτιάξει τον τρόπο εργασία μας, διαδικασίες, έχουμε ξεκινήσει, τα των ε, αντιπροσωπιών κτλ. Αλλά και εδώ είμαστε υπό εξέλιξη και θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Ωστόσο πιστεύω πως η κατάσταση τώρα είναι πολύ πιο ξεκάθαρη από ό,τι όταν ε, ξεκινήσαμε και σίγουρα είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι στην, ε, στα υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές για την οικονομική διαχείριση ε, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι πως θα ανταποκριθούμε στις ψηλότερες προδιαγραφές και στον αυστηρότερο έλεγχο και εποπτεία. Για το θέμα των προσλήψεων, ένα από τα πλεονεκτήματα της νέας δομής είναι ακριβώς ότι έχουμε το όφελος, το πλεονέκτημα μάλλον, το ότι παίρνουμε διπλωμάτες από τα κράτη-μέλη. Αυτό μας δίνει ένα νέο σύνολο ταλέντων, διαφορετικών εμπειριών, γλωσσικών, πολιτικών, αναλυτικών προσόντων και πιστεύω πως ε, πολύ καλά θα μπορέσουμε να υποφεληθούμε από όλα αυτά. Δεν θέλω να μπω στι λεπτομέρειες, αλλά ε, όταν λες ότι είναι εντυπωσιακό ότι κάποιο που μιλάει κινέζικα τώρα, στην, ε, ε, κινέζικα τώρα βρίσκεται στην Τίνιδα, δεν θέλουμε μόνο του ανθρώπου που μιλάνε κινέζικα στο Πεκίνο, πέρα από τι γλώσσε ε, χρειαζόμαστε ένα σωρό άλλα προσόντα, ένα ολόκληρο χαρτοφυλάκιο προσόντων ανάλογα με την αντιπροσωπεία που βρίσκονται και ελπίζω πω ε, πάντοτε θα μπορούμε να βρίσκουμε αυτά τα προσόντα που μπορεί να μην είναι άμεσα διαθέσιμα στο μόνιμο προσωπικό των ε, θεσμικών οργάνων. Τώρα για τα γυναίκε, αυτό η κάθε άστρο μα το θυμίζει τακτικότατα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και είναι αλήθεια, δεν είναι εξήγηση, αλλά είναι, δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι εξήγηση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και στα κράτη-μέλη ισχύει αυτή, αυτό το, η αναλογία ανδρών-γυναικών ε, και κάνουμε, σας διαβεβαιώ ότι μπορούμε. Για το θέμα των αντιπροσωπιών, το, με το υπέροχο αυτό ακρονίμιο ASAD έχουμε, που δεν ξέρω τι σημαίνει, πάντως είναι ένα σύστημα πληροφορικής που, σχεδιασμό, που, στόχο έχει να διευκολύνει την υπηρεσία μας και τις αντιπροσωπείς και τα κρατημέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Και αυτό είναι τμήμα της διαδικασίας δημιουργίας καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις αντιπροσωπείς μας, ε, ε, μάλλον στις πρεσβείες των κρατών μελών και τις αντιπροσωπείς μας. Έχουμε κάποιες δυσκολίες όπως πάντα γίνεται με τα διάφορα προγράμματα πληροφορικής αλλά είχαμε μια συνάντηση μόλι χτε γι' αυτό και ελπίζω πω έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αυξήσουμε τι δυνατότητε που έχουμε για διανομή πληροφοριών, διάδοση των πληροφοριών στα κράτη-μέλη. Υπόθηκε ότι δεν μα νοιάζει και πολύ η αναπτυξιακή πολιτική. Ε, αντίθετα πιστεύω εγώ ότι έχουμε εξάλλου κληρονομήσει ένα σωρό κόσμο που εργαζόταν στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και που είναι απόλυτα προσιλωμένη σε αυτήν την ατζέντα της ανάπτυξης. Νομίζω όμως πως ε, ξεπέρασα το χρόνο μου και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Να απαντήσω σύντομα σε κάποιε ερωτήσει. Η σημασία είναι σαφή. η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμα πολύ σημαντική χώρα όμω. Πολύ περισσότερο σε ανθρωπιστικά ζητήματα παρά σε ανάπτυξη. Και σας λέω για το τι ακούω από του συναδέλφους μου στην Αφρική και την Ασία για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Δεύτερον, για τι σε χώρες. Πάλι αυτό το οποίο μου λένε οι Ασιάτες συνάδελφοι δεν είναι μόνο ε, οι συναντήσει του υψηλότερου επίπεδου γιατί είναι περιορισμένες αλλά σε ε, όλους τους τομείς. Οι υπάλληλοι συναντώνται όλο και περισσότερο και προσαρμόζουν τις πολιτικές τους ο ένας τον άλλον και η αξιολόγηση είναι πως δεν οδηγεί σε επίσημα συμπεράσματα όπως συνηθίζουμε στην Ευρώπη αλλά σε έναν αντίκτυπο στη χάραξη της ε, πολιτικής. Για ένα άλλο θέμα της σημασία, αυτό το οποίο είπα για τη σημασία. Δεν αφορούσε μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ευρωπαϊκό μοντέλο καθεαυτό και τις ευρωπαϊκές χώρες. Το ερώτημα είναι, ε, εκλογήκαμε εμεί μετά τι εκλογέ ε, στη Βόρεια Αφρική για το ότι τόσο πολλοί άνθρωποι ψήφισαν όχι τε, πιο φιλελεύθερα αν θέλετε κόμματα αλλά ε, ε, ισλαμικά κόμματα. Δεν είναι το μοντέλο μα τόσο δημοφιλέ όσο ήταν στο παρελθόν. Αυτό είναι το θέμα. Για τις αξίε μα ναι είναι σαφές πως πρέπει να είμαστε περήφανοι που εξάγουμε τι αρχέ μα Αυτό το οποίο μου λένε όλο και περισσότερο στην συνάδελφοί μου από άλλα νότια πανεπιστήμια και διπλωμάτε ε, από αυτέ τι χώρε Είναι ωραίες οι αξίες σα, αλλά η Νότια Αφρική και η Κίνα μα δίνουν καθαρό νερό. Ε, ηλεκτρισμό. Ε, για πρώτη φορά κάποιε πόλεις του Κονγκό έχουν ηλεκτρισμό. Για ε, αυτούς. Αυτή είναι τεράστια πρόοδο. και θα ήθελαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει και τέτοια πράγματα βασικά. Και αυτό είναι σημαντικό από πλευρά νομιμοποίηση σε αυτέ τι χώρε. Πρέπει να νιώσουν πω μπορεί να έχει ένα αντίκτυπο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε κάποιες προτεραιότητες ε, τις οποίες ε, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω, όπως είπε και ο κύριος Σάλιβαν, πως ε, είχε έρθει, είπατε, πρόσωπος και στο Λουξεμβούργο, στο ελεκτικό συνέδριο και είχαμε μία ανοιχτή και ενδιαφέρουσα συζήτηση και από τις δύο πλευρές να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής σας πως είναι πάρα πολύ πιθανό πως θα κάνουμε έναν έλεγχο της υπηρεσίας αυτής, αλλά το πρόβλημα είναι πότε θα το κάνουμε. Αν δείτε ε, ε έναν τέτοιο έλεγχο θα πρέπει να γίνει πριν από το τέλος της διαδικασίας. 2014 ε, θα γίνει μια αναθεώρηση, οπότε πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ ε, τα πράγματα. Κατά την άποψή μου, ίσως μετά την αναθεώρηση η κυρία Άστον ζήτησε να ολοκληρωθεί πριν ε, ε, ολοκληρωθεί η θητεία της. Θα προσπαθήσουμε, αλλά εγώ θα πρότεινα στα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου να γίνει ένας έλεγχος πριν από το τέλος της θητείας της κυρίας Άστον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Προτείνω να ακούσουμε τώρα άλλους εννέα συναδέλφους. Το πολύ 1,5 λεπτό, αλλιώς δεν θα μιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Και η κυρία Γκρέσλε θα μιλήσει πρώτη και ξέρει καλά τα νούμερα. Παρακαλώ να προσέξει και το 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ως μια ταπεινή ελεγκτής του προπολογισμού δεν θα αναφερθώ εγώ στην εξωτερική πολιτική, να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο επιστήμονας και ε, αυτό το οποίο αναφέρεται στο σημείο 33 και 35. Έχουμε την εξής κατάσταση. Είναι η υπηρεσία αυτή πολύ χαλαρή με τον ελεύθερο χρόνο του προσωπικού της. Εάν δούμε τι γίνεται στην ΙΠΑ ε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν 8 εβδομάδες διακοπές. Ε, εδώ πέρα έχει αυτή η υπηρεσία 9, 14 κτλ. λοιπά. Κατά κανόνα είναι 25 εργάσιμες μέρες οι διακοπές. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω αυτό το πράγμα πριν το συζητήσουμε, πριν παραβιάσουμε ε, κανόνες, γιατί κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά αυτών που λείπουν, να δείτε τις διακοπές ε, της υπηρεσίας αυτής. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει λοιπόν. Δεν ετέθη το ερώτημα αυτό. Δεν θα ήθελα να χαλαρώσουν όλοι οι κανόνες χωρίς να λυθεί αυτό το πραγματικά πολύ σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Α, μα είναι, βλέπω, τόσο γενναιόδοροι όσο στη Γερμανία. Όχι, όχι, αστείευομαι, αστείευομαι. Ε, κύριε Πρόεδρε, οι Γερμανοί έχουν λιγότερες μέρες διακοπών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε. <laughs> Ναι, το, το είχα υποθέσει, το είχα υποθέσει, λέει ο κύριος Πρόεδρος. Για κονσάρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ μια μικρή χώρα και θα μιλήσω φιλανδικά. Καλό είναι να αισθάνεται κανείς ικανοποιημένος και ευτυχής και είναι πολύ ενημερωτικέ τέτοιου συναντήσεις, αλλά καλύτερο θα ήταν αν οι ε, η ΕΙΕΔ είχε μεγαλύτερη προβολή και προς τα έξω, όπως μας είπε και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Λουβά. Θα είχαμε περισσότερους λόγους για χαρά. Γιατί ε, ασκούνται τέτοιες επικρίσεις ε, προς την ΕΙΕΔ από τελευταία άτυπη συνεδρίαση γκίμικ στην Κοπεχάγη. Με βάση τον παρατηρητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν πολύ κακή εντύπωση οι ευρωπαϊκές χώρες, γιατί φαίνεται ότι είναι πιο διχασμένες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής μετά τη Λισαβόνα από ότι πριν την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Γιατί μπορεί να λέμε ότι το Παρίσι, το Λονδίνο ή ε, το Βερολίνο δεν θέλουν μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά ε, η ΑΕΔ δεν φαίνεται να επιδιώκει τη συμμαχία των μικρών χωρών που είναι η φυσιολογική εταίρη της ε, ΑΕΔ. Θα πρέπει λοιπόν ε, η ΑΕΔ όχι μόνο να προσλαμβάνει μέλη από τις μικρές χώρες αλλά και να ακούει περισσότερο τη γνώμη τους για να ενισχυθεί και η υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο κενό μεταξύ της ε, ικανοποίησης που εκφράζετε εσείς και των επικρίσεων που ακούμε από εξωτερικούς παράγοντες για την ΕΕ. Ευχαριστώ. Το κοιτάξτε, ω Γερμανός θα πω πω είναι πολιτισμένη η χρόνη διακοπών τη υπηρεσία εξωτερική δράση. Τώρα, ε, θεωρώ πώ ε, το ότι σήμερα έχουμε απαντήσει από την ε, Κομισιόν είναι κάπω περίεργο. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Λεμόν. Πρώτον. Δεύτερον, εμεί θέλουμε να έχουμε μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει ένα γενικό γραμματέα, αλλά μια ένα policy board και ένα corporate board, ένα συμβούλιο χάραξη πολιτικής και ένα συμβούλιο διοίκησης. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πότε συναντιούνται αυτές οι αρχές. Κατόπιν, για την διοίκηση. Η ευθύνη για την οικοδόμηση της υπηρεσία για εμένα ε, δεν ξέρω ποιος την έχει. Ο επικεφαλής ε, της διοίκησης είναι κάτι το οποίο ήθελε το κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε είναι πως σε αυτή τη δύσκολη φάση της δημιουργίας έχει και γεωγραφική αρμοδιότητα. Είναι κατανόητο για μένα σε τόσο πολύπλοκη ε, εποχή ο αρμόδιος για την λειτουργία. Κατόπιν, οι οδηγίες προς τις αντιπροσωπίες. Γιατί πηγαίνουν απευθείας ε, τα τηλεγραφήματα επίσης ε, στην Κομισιόν και ο κύριος Βημούν είπε πως η κυρία Άστον δεν μπορεί να βρίσκεται παντού. Εμείς το είπαμε, πρέπει να υπάρχουν πολιτικοί εκπρόσωποι της ΕΥΠΑ ΕΕ. της Ήταν η ίδια η κάθε Άστον εναντίον. Εγώ θεωρώ πως αυτό ήταν λάθος. Για μια τέτοια υπηρεσία με τέτοιο δίκτυο χρειαζόμαστε και πολιτικούς αναπληρωτές της ΕΥΠΑ ΕΕ, της Αλλιώς δεν γίνεται η δουλειά. Σας ευχαριστώ Μα το να προσκληθεί η Κομισιόν ήταν η συμφωνία των ε, κοινοβουλευτικών ομάδων. Ήταν γνωστό. Δεύτερον, η διαπίστωση σας για το πού πηγαίνουν τα τηλεγραφήματα είναι νομίζω απόδειξη για το ότι δικαίως καλέσαμε την Κομισιόν. Ε, η κυρία Κρόμπρεφ τώρα. Ευχαριστώ. Είμαι υπέρμαχο τη κοινή εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι ιδιαίτερα που η εξωτερική πολιτική έγινε πιο ρεαλιστική και πιο συνεκτική. Φυσικά χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμό και ε, ηγετικό ρόλο σε θέματα εξωτερικά, αλλά είμαστε στη σωστή πορεία. Η κυρία Κονσάρη μίλησε για τη διχασμό που παρατηρείται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και την επιρροή που έχουν οι μικρές χώρες στη διαμόρφωση τη εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι μόνο θέμα προσωπικού της ΕΙΕΔ, είναι και θέμα εκπεριτροπής προεδρίας, κάτι που δίνει ενάψματα στις μικρές χώρες για περισσότερη ενεργοποίηση, να, για να ακουστεί η φωνή τους και ίσως ε, η εκπεριτροπής προεδρία είναι ο καλύτερος τρόπος για να κινητοποιήσουμε τις μικρές χώρες που στο παρελθόν ε, είχαν μπει στο, παρασκήνιο από τις ε, μεγάλες χώρες που μονοπόλησαν την εξωτερική πολιτική. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε πριν από εννέα ομιλητές ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι σημαίνει σημαντική πρόοδος στην περίπτωση αυτή. Σημαντική πρόοδος στην ε, δαπάνη κονδυλίων και στην σελίδα 16 της έκθεσης έχουμε μια καταθλιπτική ε, διατύπωση για διαρθρωτικό έλλειμμα, που σημαίνει ότι ακόμη περισσότερα κονδύλια θα δαπανηθούν. Αναφέρθηκε προηγουμένως η Λιβύη και ε, θα ήθελα να πω ότι έχουμε 27 χώρες μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξι ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν ε, στην στο συνασπισμό κατά του καθεστώτος Καντάφη και μόνο τέσσερις από τις έξι χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κοινή θέση για θέματα εξωτερικής πολιτικής, για σημαντικά ζητήματα. Δεν υπάρχει καν κοινή εξωτερική πολιτική. Και ολόκληρη η ΑΕΔ στηρίζεται σε έναν μύθο εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκή πολιτεία, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι αντικείμενο άλλη συζήτηση. Αναφέρθηκε ότι η ΕΕΔ εκπροσωπείται με πολυμερή αντιπροσωπεία στα Μπαρμπάντος. Ε, καθόλου περίεργο. Φαίνεται ότι έχουν, είναι, πολιτισ, είναι ε, επιτετραμένοι για πολιτιστικά θέματα. Δεν ξέρω αν ε, η πρόταση για τους ε, επιτετραμένους γεωπολιτιστικά θέματα είναι μια πρόταση που θα ευοδοθεί. The floor has, sorry, Mr. Thank you, uh, Chairman. General remark. I think that EAS is. Uh... Κύριε Πρόεδρε, μια γενική παρατηρήση. Η υπηρεσία αυτή είναι ένα μέσο και όχι αυτός ο σκοπός. Το πρώτο μου ερώτημα είναι πως υπάρχει ένα κενό και μία αντίθεση μεταξύ της πολύ θετική αυτοαξιολόγησης ε, από την υπηρεσία και των επικρίσεων από όποιον είναι έξω από την υπηρεσία. Το ερώτημα είναι γιατί. Δεύτερον, για τις προσδοκίες της ψηλές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για γεωγραφική υπηρεσία και ισορροπία και ισορροπία των δύο φίλων. Στο δε σημείο 26 της ε, έκθεσης της ΥΠΑ της εκπροσώπου λέει πως σημειώθηκε καλή πρόοδος δεν αρκεί αυτό. Δεν υπάρχει ε, πρόοδος και υπάρχει μεγάλη ανισορροπία. Αν συνεχιστεί αυτή η αυτοικανοποίηση της υπηρεσίας, τα διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν το 2013. Τρίτο μου ερώτημα. Ε, θεωρείτε πως έχει υπάρξει κάποια επίδραση της κρίσης και αλλαγή άρα του... της εστίασής σας. Κατόπιν, πόσο ικανοποιημένοι είστε με τις προτάσεις του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ή μήπως θα δούμε όπως λέγαμε πάντα εδώ πέρα πως η εξωτερική πολιτική της Ένωσης είναι ε, υποχρηματοδοτούμενη. Και τελευταίο ερώτημα, αφού είμαστε τόσο ικανοποιημένοι γιατί χάνουμε το μέτωπο της ανατολικής μας ε, γειτονίας. Σας ευχαριστώ. Κύριε, Κύριε Χάουιτ, ε, εγώ θα αγνοήσω αυτό το σχολιάκι για Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ε, για να μην πω και ο συνάδελφο, πως δεν είμαι αρκετά Βρετανός. Λοιπόν, ε, Άλντε, σοσιαλιστέ και ΕΛΚ αξιολόγησαν θετικά την υπηρεσία. Πρέπει να το πω, οι εθνικοί υπάλληλοι που πήγαν εκεί πέρα έχουν ενσωματωθεί πάρα πολύ καλά και συμφωνώ με τον κύριο Τάνοκ πως ε, οι διορισμοί ήταν εξαιρετικοί. Και όσον αφορά τις ελλείψεις, η εντολή να μην αναλαμβάνουν ρίσκο είναι εντολή του Συμβουλίου. Εάν θέλουν περισσότερο ρίσκο αυτό πρέπει να αποφασίσουν. Πιο ερωτήσει προ προς κυρίου Βημό ή ο Σάλιβαν. Μιλήσαμε για την Αραβική Άνοιξη, νομίζω πως πρόκειται για ε, επίδεγμα. Ε, θέλετε να μας δώσετε παραδείγματα άλλων χωρών όπου βλέπετε κάποιο επίδεγμα για τον ε, κύριο Σεύκοβιτ, τον κύριο Επίτροπο. Γιατί υπάρχει περισσότερο προσωπικό της ε, Επιτροπής ε, από της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ένα χρόνο μετά. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Για το ελεγκτικό συνέδριο, όταν εξετάζετε τις δαπάνες ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, λαμβάνετε υπόψη το έργο της προηγούμενης Προεδρίας όταν είχαμε Προεδρίες με το επιχείρημα αυτό το ψεύτικο της ουδετερότητας ε, του υπερπολογισμού. Ε, Προ τον κύριο από το Κολέγιο τη Ευρώπη, ε, εγώ, επειδή εγώ έχω πάει στην αντιπροσωπεία του Βερολίνου, το να λέτε ότι δεν μιλάει κανεί Κινέζικα είναι απλά λάθο. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι εκεί πέρα. Αν θέλετε περισσότερου ειδικού, πού θεωρείτε εσεί ότι, από πού θεωρείτε ότι θα πρέπει να προέλθουν. Πρόεδρε, Ο Πιέρ είπε Όταν ξεκινήσαμε την απόψινή συνεδρίαση, πως τα κράτη-μέλη είχαν την φιλοδοξία για μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια. Ξέρουμε ότι δεν επιθυμούν ε, από την ΕΙΕΔ. Ίσως θα μπορούσαμε να ακούσουμε τι πιστεύουν πως επιθυμούν από την ΕΕ τα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο. Εάν δεν το ορίσουμε αυτό, θα είναι προβληματικό στο να ξεκινήσουμε μια σοβαρή ε, θεώρηση αυτή της υπηρεσία την οποία έχουμε προγραμματίσει για το 2013. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι πόσο εκτεταμένη πιστεύετε ότι μπορεί να είναι μια τέτοια αναθεώρηση. Μπορούμε εκ νέου να εξετάσουμε το θέμα των πολιτικών εντεταλμένων, της ε, ε, επιχειρησιακής δομής διαχείρισης και τις δυνατότητες προγραμματισμού. Όσον αφορά την ομάδα μου, εμείς θα θέλαμε να γίνει μία ε, πανεξέταση των φιλοδοξιών. Εν γέννη είμαστε όμως ικανοποιημένοι, όπως και κάποιοι άλλοι ομιλητές, από την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής. Danke, Herr Vorsitzender. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα αναφερθώ στο ερώτημα του κυρίου Κόγκελε. Ποια είναι η σημασία της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Και εδώ πέρα θα ήθελα να σας παρακαλέσω εάν ε, παρατηρήσατε τι γίνεται με την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνος περιφερειακός οργανισμός που έχει τέτοια πολιτική. Μπορέσατε να παρατηρήσετε τυχόν αποτελέσματα και στις χώρες Μπρίκ αλλά και πολυμερός. Και το ίδιο ερώτημα θα ήθελα να απευθύνω και στον κύριο Βημό. Τι αξιολόγηση έχουν κάνει στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων επισημάθηκε κυρίως το θέμα της αποδοχής της ΑΕΔ από τα κράτη-μέλη. Σίγουρα η αρχή ήταν δύσκολη και χρειάστηκε και μια αλλαγή νοοτροπίας ορισμένων χωρών μελών και υπουργών εξωτερικών. Αλλά και εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για κάθε κράτος μέλος. Πάντως μπορούμε επιτέλους να δείξουμε ε, πόσο σημαντική είναι η συνεργασία και τι προστιθέμενη αξία υπάρχει και πόσο πιο σημαντική γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν καταφέρνει και αποφαίνεται με ενιαία φωνή και πόσο μεγαλώνει το βάρος της στην εξωτερική πολιτική όταν έχει μία διάσπαστη φωνή στο G20, στο G8 ή σε άλλες σημαντικές ε, διεθνείς διασκέψεις κορυφής. Φαίνεται τότε η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι πιστικά αυτά τα επιχειρήματα, ακόμη και για τις χώρες που αρχικά ήταν κάπως επιφυλακτικές για τις εξελίξεις και την πορεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ό,τι αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων, την ενημέρωση ε, της Επιτροπής και τις σχέσεις Επιτροπής ΑΕΔ. Όπως είπε και ο κύριος Σάλιβαν, αυτά τα θέματα συζητήθηκαν αλλά και διευθετήθηκαν. Έχουμε κάποιες κοινέ δομές, έχουμε κοινό προσωπικό σε αντιπροσωπείες και όταν λέμε για οδηγίες από τις ε, επιμέρους ε, γενικές διευθύνσεις προς τους ε, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Ε, ενημερώνεται η ΕΕΔ, ενημερώνεται ο επικεφαλή Αντιπροσωπεία και το ίδιο ισχύει και για την αποστολή των ε, εκθέσεων από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Πηγαίνει στον, πηγαίνουν στον πρέσβη, στην αρμόδια γενική διεύθυνση, αλλά στέλνετε αντίγραφο και στην ΕΙΕΔ ΕΕ αυτών των εκθέσεων. Δεν υπάρχει πια πρόβλημα. Τώρα ως προς τον προϋπολογισμό. Φαντάζομαι θα σχολιάσουν το θέμα αυτό και οι συνάδελφοι από την ΕΙΕΔ. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι θέτουμε πολύ ρεαλιστικές προτάσεις για, τον, για το κεφάλαιο 5. Στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις στο Συμβούλιο τα πράγματα δεν ήταν εύκολα και γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι ακαθόδεις. Πάντως, εμείς υποβάλαμε προτάσεις με σημαντικές περικοπές και φυσικά θέλουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας. Πάντως ε, πιστεύω ότι η πρόταση που καταθέσαμε είναι λειτουργική, γιατί θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε ε, μια εύρυθμη λειτουργία της ΕΙΕΔ προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Και ελπίζω ότι η πρόταση θα υποστηριχθεί και από το Κοινοβούλιο και αργότερα από το Συμβούλιο. Τώρα, γιατί έχουμε περισσότερους υπαλλήλους της Κομισιόν στις αντιπροσωπείες από ό,τι εμπειρογνώμονες της ΕΙΕΔ. Είναι φυσικό κάτι τέτοιο. Είναι λογικό γιατί οι υπάλληλοι της ε, Κομισιόν είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου, που είναι περίπου 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε την ευθύνη απέναντι στην αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή να χρησιμοποιούμε σωστά αυτά τα κονδύλια. Λογικά και με χρηστή διαχείριση. Οπότε σχεδόν αποκλειστικά οι υπάλληλοι της Κομισιόν στις αντιπροσωπείες είναι οι υπάλληλοι της ΔΕΦΚΟ και οι υπόλοιποι είναι υπάλληλοι της Κομισιόν. Οπότε ε, προσωπικό της ΕΙΕΔ είναι τοπική πάλι. Γι' αυτό και ε, είναι τόσο σημαντική η παρουσία των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ε, αντιπροσωπείες ανά τον κόσμο. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. δεχτήκαμε κριτικές ότι είμαστε πολύ διχασμένοι στο γκίμιχ. Ε, δεν ε, είχαμε αυτή την αίσθηση. Μάλιστα, οι περισσότεροι υπουργοί που ήρθαν ε, θεώρησαν αντίθετα πως είχαν πολύ πιο περισσότερα κοινά από ό,τι είχαν ε, παλιότερα. Και το, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ίσως θα πρέπει να γίνει καλύτερη αξιολόγηση του τι ακριβώς συνέβη στο γκίμνηση. Τώρα, το θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας. Συμφωνώ πως αυτό είναι πρόβλημα για πολλά από τα κράτη-μέλη που πιστεύουν πως κάτι έχασαν εκεί. Και νομίζω πως είναι πρόβλημα για την ΑΕΔ να προσπαθεί να διατηρεί διαρκώς ε, την ε, όθηση στην ΚΕΠΑ, ε, ενώ η Προεδρία η περιτροπή είχε ένα διάστημα εξάμεινο που μπορούσε να πολύ ενέργεια να ε, χρησιμοποιήσει, ενώ εμείς πρέπει να διατηρούμε αυτή την ενέργεια για μονίμως. Για την εκπεριτροπή τη Προεδρίας βεβαίως η ΕΔΕ δεν έχει αλλάξει τον κόσμο, αλλά είμαστε ειλικρινεί. Θα πρέπει να δούμε ότι αυτό οφείλεται και στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού, στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ήταν η ναυαρχίδα ε, αυτής της εργασίας και το έχουν χάσει τώρα αυτό και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα τη Λιβύη Είπαμε ότι έξι στην ουσία τέσσερα μόνο καδημέλη ε, ε, πλάκησαν στις στρατιωτικές, στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η πολιτική στάση που κράτησε η Ευρώπη ήταν απόλυτα ενωμένη και ήταν εντυπωσιακή μάλιστα σε σύγκριση με τις ε, διαφορές που είχαμε σε σχέση με τη στατιωτική επιχείρηση. Σκεφτείτε μισό λεπτό τον τρόπο με τον οποίο τα 27 κατημέλη αρκετά γρήγορα κατάφεραν να συμφωνήσουν για τον τρόπο που θα έπρεπε να ενεργήσουν σε σχέση με το ε, παραδοσιακό Εθνικό Συμβούλιο στη Βενγάζη. Όλοι πήγαν στη Βενγάζη για να στηρίξουν αυτές τις νέες αρχές που αναδύονταν και το γεγονός ότι καταφέραμε αρκετά ομαλά και γρήγορα να παρουσιάσουμε κοινό μέτωπο και να ενεργήσουμε από κοινού απέναντι στη Λιβύη. Πρέπει κανείς να το θυμάται αυτό. Ε, Επίση ρωτήθηκε και είναι πολύ καλή ερώτηση. Βέβαια δεν είμαι σίγουρο ότι έχω τη σωστή απάντηση. Αλλά θα δοκιμάσω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στι επικρίσεις που δεχόμαστε εκτός ε, από κάποια δεξαμενές σκέψεις τα think tanks και των όσων οι ίδιοι επικρίνουμε στους εαυτούς μας. Εγώ νομίζω πως είμαστε αρκετά πιο ταπεινοί. Ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε πολλά, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και ε, δυσκολίες και ότι ακόμα έχουμε μεγάλο έργο μπροστά μας, αλλά με εντυπωσιάζει και το γεγονός ότι τα Αυτές οι δεξαμενές που βασίζονται, που εδράζουν στις Βρυξέλλες ε, ήταν πολύ επικριτικές, ενώ άνθρωποι εκτός των Βρυξελών ε, υποστήριξαν πολύ περισσότερο τα όσα προσπαθούμε να κάνουμε. Και τρίτες χώρες που επανειλημμένως έρχονται στις Βρυξέλλες να μας επισκεφθούν, φαίνεται να είναι πολύ πιο ευχαριστημένοι με τον τρόπο που προσπαθούμε να δουλέψουμε από ότι θα ακούμε και διαβάζουμε στις εκθέσεις εδώ. Με ρωτήσατε αν είχαμε άλλες επιτυχίες εκτός από τις χώρες τη Αραβικής Άνοιξη, χωρί να ε, θέλω να αυτοεπαίρνουμε. θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια πράγματα. Σαχέλ, Σομαλία, Κέρας Αφρικής, ακόμα και αναδυόμενες χώρες όπω η Βραζιλία. Τα πάμε πάρα πολύ καλά με τη Βραζιλία. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με τη Βραζιλία. Τέλος, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα το τι σημασία έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για την Αιέδη στην Αφρική, για παράδειγμα. Να σας αναφέρω απλά πώς προχωρούμε με την υπόθεση των αποστολών παρακολούθηση των εκλογών. Η Τινησία μας ζητά, η Αλγερία μας ζητά, η Λιβύη μας ζητά τεχνική βοήθεια ε, σε αυτό το τομέα και νομίζω πως αυτό είναι καλό ε, μήνυμα για το τι μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Οσάλιβαν. Σύντομα. Γιατί ξέρω πως ο χρόνος πιέζει. Πρώτα απ' όλα ελπίζω να μην ε, θεωρείτε πως ε, παριστάνουμε τους έξυπνους ή έχουμε ε, χαλαρώσει. Ε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά το τι πρέπει ακόμα να γίνει για να ε, στηθεί ο οργανισμός μας. Απλά προσπαθώ να πω πως έχουμε επιτύχει κάποια πρόοδο από όταν ξεκινήσαμε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και θα σας υπενθυμίσω πως η φύση της υπηρεσίας είναι να συγκεράσει προσωπικό της Κομισιόν, της Γραμματείας του Συμβουλίου, των αντιπροσωπείων, πράγματα τα οποία υπήρχαν, πληρώνονταν και ελπίζουμε να προσθέσουμε κάποια αξία και ε, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί καμιά φορά υπάρχει εντύπωση που δημιουργούμε κάτι το τελείω καινούριο. Ε, Εμεί ελπίζουμε απλά να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό για το ζήτημα των διακοπών, που δεν είναι αμεληταίο. Συμφωνούμε με την κυρία Γκρέσλε. Πράγματι, ε, σε γενικές γραμμές δεν ε, είμαστε στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις άδειες του προσωπικού που για διάφορους λόγους ε, είναι υπερβολικές. Για τις ε, οδηγίες προς τις αντιπροσωπείες που ανέφερε ο κύριος Λάμπστορφ απάντησε ο αντιπρόεδρος ο κύριος Σεύκοβιτς. Εγώ ήμουν γενικός διευθυντής εμπορίου στην Κομισιόν, έστελνα οδηγίες στις αντιπροσωπίες Δεν νομίζω πως υπάρχει πρόβλημα για το ερώτημα του κυρίου Σάριου Βόλσκι για τη γεωγραφική ισορροπία. Δέχομαι πως δεν μπορέσαμε να διορθώσουμε την κατάσταση όσο θα θέλαμε. Να θυμάστε πως ξεκινήσαμε με το προσωπικό που είχαμε, που ούτως ή άλλως δεν είναι αντιπροσωπευτικό όλων των κρατών μελών. Αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο με την εισρωή, που είναι ούτως ή άλλως ε, λίγων θέσεων. Αλλά η κάθε άστον είναι υπέρ και αν δείτε την ανάλυση των νέων προσλήψεων. Νομίζω πως σιγά σιγά σημειώνουμε πρόοδο, αλλά δέχομαι πως αν δείτε την ανισορροπία πράγματι δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση. Για το θέμα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου είμαστε ικανοποιημένοι με τις προτάσεις της Κομισιόν για νέα εξωτερικά μέσα. Η Κομισιόν έχει προτείνει αύξηση στην εξωτερική χρηματοδότηση. Αυτό νομίζω δικαιολογείται ε, ζητάμε στήριξη από το Κοινοβούλιο στις δύσκολες συζητήσεις που θα ακολουθήσουν και ελπίζω να το δούμε τον ίδιο τρόπο και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ρώτησα ποιο ήταν ε, το προβλεπόμενο εύρος και η φύση ε, της αναθεώρησης του 2013. Δεν ξέρω αν ο κύριος Βιγιόμ ή ο κύριος Σάλιβαν ε, θα ήθελαν να απαντήσουν αυτή την ερώτηση. Νομίζω, ε, εάν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, νομίζω κύριε Ντάφ πως είναι ανοιχτό το ζήτημα και οπωσδήποτε είπα ότι εκπρόσωπος ε, δεν έχει τοποθετηθεί από όσο ξέρω. Το ερώτημα θα πρέπει να συζητηθεί ε, θα έχετε ζήσει και εσείς και άλλοι τις δυσκολίες δημιουργίας της υπηρεσίας είναι πολιτικό το ζήτημα, πόσο θέλουμε να ξανανοίξουμε τα δύσκολα αυτά ερωτήματα, ακόμα και αν εκ των υστέρων βεβαίως ε, θεωρούμε πως μπορούσαν να γίνει κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Για μένα το ζήτημα είναι το να σπαταλάμε ενέργεια και πολιτικό κεφάλαιο και να μην έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά ειλικρινά σας λέω πως θεωρώ πως είναι ανοιχτό το ερώτημα και οπωσδήποτε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα αποφασίσουν σε ποιο βαθμό θα προχωρήσει η θεώρηση. Εμείς τώρα μόλις ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε πώς θα δώσουμε τα στοιχεία που θα ζητήσει η ύπατη εκπρόσωπος και θα είναι πολιτική επιλογή το σε ποιο βαθμό θα ξανανοίξουμε ζητήματα που έχουν ήδη κλείσει σε νομικά ζητήματα. Αλλά σας υπενθυμίζω πως ήταν πάρα πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις ε, πριν ε, από 18 μήνες. Δεν είναι πολύ ικανοποιητική απάντηση, μόνο αυτή όμως μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις του κ. Χόουιτ, είναι πολύ πιθανό ότι θα γίνει λογιστικό έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Και είπα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει τέτοιο λογιστικό έλεγχο για θέματα όπως αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, οικονομία, εξοικονομήσεις. Βέβαια δεν μπορούν όλα να γίνουν ταυτόχρονα και ε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε στοχευμένους ε, ελέγχους. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα είναι σίγουρα γιατί ε, θα είναι λογιστικός για τα, για τα κονδύλια που έχουν ε, δαπανηθεί. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να χαρακτηρίσουμε το είδος του ελέγχου και σε ποιο τομέα θα αναφέρεται. Μία σύντομη απάντηση στις ερωτήσεις του κ. Χάουιτ και της κυρίας Λόχμπιλερ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βρετανοί συνάδελφοι κυρίω στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και ο συνάδελφος Καλπνίθ είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλο και πιο συνεπής και συνεκτική στην πολιτική τη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θετική αυτή η εξέλιξη. Βέβαια, φαίνεται ότι και οι δύο εμπειρογνώμονε διαπίστωσαν ότι ε, για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται ότι ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο συνεπής, αλλά φαίνεται πιο απομονωμένη. Στα Ηνωμένα Έθνη οι υπόλοιπε χώρες δεν φαίνεται να την ακολουθούν. Ακόμη και η Βραζιλία, η Νότια Αφρική που είναι δημοκρατικές χώρες φαίνεται ότι δεν ακολουθούν την, Πολιτική Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράδοξο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διευρύνουμε την προοπτική μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι συνάδελφοι προτιμούν βέβαια να έχουν καθαρό νερό πόσιμο είδωρ στις πόλεις τους, γιατί έτσι μεγαλώνει το προσδόκιμο ζωής από τα 49 ίσως το 57 έτη. Οπότε αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντικά τέτοιου, τέτοιου είδους στοιχεία. Τώρα σε ό,τι αφορά την Κίνα και τη γνώση των Κινέζικων. Στο, στο Πεκίνο λίγοι στην αντιπροσωπεία μιλούν Κινέζικα. Δεδομένως όμως της ε, τεράστιας σημασίας της Κίνας, ρωτώ, έχουμε αρκετούς που μιλούν άπτεστα κινέζικα και μπορούν να έχουν επαφές ε, ε, ή να παρακολουθούν τις εξελίξεις από πρώτο χέρι. Δεν νομίζω. Το θέμα των εμπειρογνώμων είναι πολύ δύσκολο δεν έχουμε τέτοιες ε, παραδόσεις όπως έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου οι σπουδαστέ, ε, είναι υποχρεωμένοι να μαθαίνουν αραβικά, κινέζικα ή ρωσικά. Στις ευρωπαϊκές σπουδές ε, έχουμε περισσότερο, δίνουμε περισσότερη έμβαση στις αφρικανικές χώρες παρά στις ασιατικές. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι όλο και περισσότεροι άλλο θα πει εκτός Ευρωπαϊκής από την Κίνα, την Κορέα, την Αφρική εργάζονται ε, σε αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κορέα αλλού ή συνεργάζονται με, ε, στα γραφεία των Ευρωβουλευτών. Νομίζω ότι μπορούμε να ε, υποστηρίξουμε τέτοιο κλάδο σπουδών, την ανάπτυξη τέτοιου κλάδου σπουδών στο μέλλον και φυσικά να δίνουμε έμφαση στην ανταλλαγή φοιτητών ε, και να επιτρέπουμε σε φοιτητέ να έρχονται και να εργάζονται από τι χώρε αυτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για το ότι ήρθατε, μας μιλήσετε και απαντήσατε σε ερωτήσεις. Βεβαίως η συζήτηση αφορούσε την λειτουργία της ε, υπηρεσία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Κατ' ξεκίνησε η υπηρεσία να λειτουργεί Δεκέμβριο 2010, πριν 14-15 μήνες. Δεν μπορεί να είναι τα πάντα τέλεια, αλλά πρέπει να δούμε το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να γίνει καλύτερη αυτή η υπηρεσία και που έχουν γίνει λάθη, γιατί νομίζω αυτός είναι ο κοινός μας στόχος. Να έχουμε μια καλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο καλής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλής. Και, γράφει η κυρία Γκρέσλε εδώ πέρα, σε λογική τιμή. Νομίζω ακούσαμε κάποια πράγματα. Μπορεί να διαβάσει κανείς τα πρακτικά μετά αυτής της ακρόασης και να βγάλει τα συμπεράσματά του με τρόπο πιο συστηματικό να συζητηθούν τα αυτά και έτσι να βοηθήσουμε και ταυτόχρονα στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση ε, του 2013 να, να προετοιμαστούμε. Και ο Σπίνγκστεν, ε, αν και βεβαίως δεν υπήρξε πλήρης έλεγχος, μας ε, έδωσε κάποιες ενδείξεις οι οποίες οπωσδήποτε βοηθούν. Για να μην πηγαίνουμε σε λάθος κατεύθυνση. Θεωρώ πως ναι, ήταν καλή αυτή η ακρόαση. Και αναφέραμε και το ζήτημα της συνεργασίας με την Κομισιόν. Γιατί υπήρχαν κάποια προβληματάκια, τώρα φαίνεται πάνε καλύτερα τα πράγματα. Θα βρεθούμε βεβαίω και σε αντιπροσωπείες, θα δούμε τι γίνεται στην πράξη. Γιατί βεβαίω ε, έχουμε και ανθρώπους που στελεχώνουν αυτές τις θέσεις και θεωρώ πως η δυσκολία είναι πως το πολιτικό κομμάτι των αντιπροσωπιών και για λόγους ιστορικούς πάντα ήταν πολιτική εμπορίου και αναπτυξιακή και τώρα υπάρχει μια πολιτική διάσταση για να γίνει μια πλήρης εξωτερική υπηρεσία. Και οπωσδήποτε θα χρειαστεί κάποια ώρα. εκεί πέρα θα έχουμε τα ωφέλη της συνέργειας για τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής. γιατί βεβαίως ε, έτσι θα μπορεί με τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η να διαμορφώσει μια τέτοια πολιτική. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δούμε και τις συμφωνίες που έχουμε κάνει και σχετίζονται με λογοδοσία και τα σχετικά. Έχω την αίσθηση πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. και θα πρέπει να υπάρξει και ο έλεγχος, αλλά να μην ε, εμποδίζει, νομίζω. Αλλά να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος οπωσδήποτε. Και θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός εδώ πέρα. Θα γίνει λοιπόν αυτό και θέλω να σας παρακαλέσω να είστε εκεί στην ε, διάθεσή μας για να έχουμε έτσι μια βάση για μέση συζήτηση για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ορίστε. Ναι. Ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Καλό σας βράδυ.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε την μεγάλη χαρά να υποδεχτούμε στη συνεδρίασή μας τον κύριο Μάρτιν Κόμπλερ. Χαίρομαι ιδιαίτερο για την συμμετοχή του στη συνεδρίασή μας και παρά τις δυσκολίες βρήκε χρόνο στο πρόγραμμά του για να μας επισκεφτεί. Μας χαροποιεί ιδιαίτερο αυτό. Έχουμε και τον κύριο Μινέλη. Μιγκαρέλη, Μιγκαρέλη συγγνώμη, το Γενικό Διευθυντή ε, της ε, ΑΕΔ ε, για τα θέματα του Ιράκ. Θα γίνει μια ενημέρωση. Ελπίζω να είναι καλές οι ειδήσει, γιατί υπάρχουν δίσταμες μέσα ιδιαίτερα στο τη φορά το στρατόπεδο ΑΣΑΦ. Ο Μάριο Μάουρο είναι ο εισηγητής μας για το Ιράκ. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Κόμπλερ για να μας εξηγήσει την κατάσταση στο Ιράκ και μετά θα γίνει συζήτηση. Κύριε Κόμπλερ, έχετε το λόγο. Ε, μεγάλη μου τιμή και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Θα ήθελα να ξεκινήσω με, με κάποιες γενικές παρατηρήσεις για το Ιράκ, αν θέλετε κι εσείς, να μην εστιάσω την προσοχή μόνο στο Ασράφ. Μόλις έρχομαι από τη Βαγδάτη, έφτασα σήμερα το πρωί και χθε είχαμε μια πολύ δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά την βία που προκάλεσε 50 θύματα και εκατοντάδες τραυματίες. Βέβαια, φανταστείτε ότι αυτό είναι πολύ καλύτερο από ότι το 2006 και το 2007. Ωστόσο, κάθε άνθρωπος, γυναίκα, παιδί που πεθαίνει στους δρόμους του Ιράκ περισσεύει πια. Δεν είναι θέμα στατιστικής, αλλά αποδεικνύει απλά ότι η κατάσταση είναι καλύτερη από ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Ωστόσο, υπάρχει τεράστιο ε, δυναμικό δρομοκρατικών δραστηριοτήτων, ομάδων που χρησιμοποιούν τη βία για να ε, επιτύχουν τους πολιτικούς τους στόχου. Τώρα, σε τι οφείλεται αυτό οι λόγοι είναι πολλαπλοί. Ένας είναι η έλλειψη της πολιτικής διαδικασίας, η έλλειψη συμπεριλήψης όλων των τριών συνιστοσών, πολιτικό τέλμα, όλοι περιμένουν ε, μια εθνική διάσκεψη ώστε οι πολιτικές δυνάμεις να συγκεντρωθούν. Ε, ένας άλλος λόγος είναι και η περιφερειακή δυναμική φυσικά, γιατί το Ιράκ είναι μια χώρα που γεωστατηγικά βρίσκεται στη μέση ανάμεσα στη Συρία και τα προβλήματά της και το Ιράν με το Κουβέιτ νότια που δεν έχει τελειώσει εκεί η υπόθεση. Και αυτό που κάνουμε από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών είναι να παρεμβαίνουμε εδώ, όχι να παρεμβαίνουμε, να βοηθούμε μέσα στο πλαίσιο της εντολής μας που δεν είναι και εντολή κεφαλαίο 7, είναι κεφάλαιο 6 η εντολή μας μετά από το αίτημα της κυβέρνησης με έργο να προωθήσουμε την εθνική συμφιλίωση, να συγκεντρώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις και εδώ αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Ε, το θετικό είναι ότι Είχαμε, έχουμε την διάσκεψη κορυφής της Αραβικής Ένωσης, ε, μεγάλο βήμα, Βαγδάτη, οι Ιρακινοί άφησαν την Προεδρία συγγνώμη, θα έχουν την Προεδρία για ένα έτος, πράγμα που θα δημιουργήσει μια πολιτική δυναμική που μας κάνει να ελπίζουμε. Όμως υπάρχουν κάποια εκκρεμή προβλήματα με τον Κουβέιτ, ο Πρωθυπουργό ε, πήγε στο Κουβέιτ, υπήρξε πρόοδος, όμως υπάρχει ε, η ολοκλήρωση του κεφαλαίου 7 που πρέπει να ολοκληρωθεί, είναι 70 δις ε, δολάρια που εκκρεμούν και που πρέπει να καταβληθούν στο Κουβέιτ αλλά και εκεί φαίνεται να υπάρχει πρόοδος και να θέλουν να γρήγορα να ολοκληρώσουν το θέμα αλλά είναι ψυχολογικό το θέμα. Δεν θέλουμε εμείς να πληρώσουμε για τις αμαρτίες των ε, ε, προγόνων μας. Θέλουμε να φύγουμε από το κεφάλαιο 7. Αυτό είναι το συνοριακό πρόβλημα με το Κουβέιτ και το θέμα της αποζημίωσης. Πρόβλημα συνόρων μάλλον. Τουρκία το βορρά, Κουβέιτ στο νότο, Ιράν προς Ανατολάς και Συρία προς Δυσμάς. Ε, εκεί βρίσκεται το Ιράκ. Και όπως καταλαβαίνετε η περιφερειακή δυναμική είναι πολύ δύσκολη. Στο Ιράκ, 8 χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, έχουν πολλά θέματα μείνει σε κρεμότητα, ιδιαίτερα στο πολιτικό τομέα. Πολλέ ε, συνταγματικέ διατάξει δεν έχουν υλοποιηθεί. Αυτό συμβαίνει με το δεύτερο σώμα, δηλαδή το Συμβούλιο τη Ομοσπονδία, η νομοθεσία περί μειονοτήτων και προστασία αυτών, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα σωρό άλλα. Και αυτό που περιμένει ο λαός του Ιράκ και εδώ πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε γι' αυτό είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η καταπολέμηση της ευθοράς, κράτος δικαίου, ο σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και α, παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα. Και ε, εστιάζεται η προσοχή στην πολιτική διαδικασία, αλλά τα αιτήματα του λαού ε, να φροντίσουν δηλαδή τις δικέ τους ανάγκε. όσον αφορά την παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα, όπω ο ηλεκτρισμό, παροχή ηλεκτρισμού για παράδειγμα, δεν γίνονται πολλά. Και το ίδιο συμβαίνει και για την παιδεία. Να πω δύο λόγια για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας. Εδώ θα εκμεταλλευτώ το ότι έχω το λόγο και σας απευθύνω αυτά τα λόγια. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ισχυρή πολιτική εκπροσώπηση στο Ιράκ. Όπως σας περιέγραψα, το Ιράκ δεν θα πρέπει να ξεχαστεί. Είναι ε, γεωστρατηγική σημασία η χώρα αυτή ανάμεσα στην Τουρκία, το Κουβέιτ, το Ιράν και τη Συρία με πολλούς ε, ενδιαφερόμενους που ενδρούν στη χώρα. Τα Ηνωμένα Έθνη και μάλιστα μέσα στη δική μας εντολή είμαστε μόνος διεθνής οργανισμός που έχει απομείνει μετά από την Αμερικανική απόσυρση στα τέλη του περασμένου έτους η χώρα είναι απόλυτα κυρίαρχη με το δικό της στρατό, με τη δικά της πολιτικά προβλήματα και χρειάζεται στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η... Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύεται εκεί από μια πολύ δραστήρια και φιλόδοξη φιλόδοξο μάλλον ε, πρέσβη εκεί, με έχουμε, με την οποία έχουμε πολύ στενές σχέσεις. Ωστόσο, ο χώρος όπου ζει δεν είναι ο ιδανικός και αυτό εμποδίζει την εκπροσώπηση της Ένωσης δεν μπορεί να, δηλαδή να αναπτύξει ένα είδο δημόσια εικόνας μέσα στο πλαίσιο των Ιρακινών αρχών. Συχνά τα κράτη-μέλη θέλουν να περιορίσουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θέλουν να περιορίσουν το ρόλο των εθνικών πρεσβειών σε έναν οικονομικό απλά ρόλο. Ωστόσο εμείς, ε, ο ΙΕ, έχουμε ειδικά πολιτικές ε, αποστολέ και δεν θέλουμε αυτό να το κάνουμε από μόνοι μα μεμονωμένα. Θέλουμε τη στήριξη των υπολείπων είτε είναι πρεσβείες είτε οτιδήποτε άλλο και πάνω απ' όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό και ε, θέλουμε να έχει χρειάζεται ισχυρή πολιτική εκπροσώπηση ξέρω βέβαια του οικονομικές, τους οικονομικούς περιορισμούς και των κρατών μελών αλλά και της Ένωσης Ωστόσο θα πρέπει να εκπροσωπηθούν με πιο ισχυρό τρόπο. Έχουμε λοιπόν εγχώρια και πολιτικά προβλήματα από τη μια πλευρά, εκρεμή ζητήματα που δεν περιορίζονται μόνο στα συνταγματικά ζητήματα αλλά και σε πρακτικά προβλήματα όπως το νομοσχέδιο για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αλλά αυτό το νομοσχέδιο εκρεμεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Είναι πλούσια χώρα το Ιράκ και αυτό πρέπει να περάσει. Γιατί θα δώσει ασφάλεια για επενδύσει, θα δώσει ασφάλεια για τι θέσει απασχόληση. Και όλα αυτά είναι προσπάθειε που εμεί μόνο και κάποιε διμερεί πρεσβείε δεν μπορούν να ε, στηρίξουν. Πολιτικές εξελίξεις αλλά και οικονομική ατζέντα της χώρας θα πρέπει να προχωρήσει προς όφελος του λαού του Ιράκ. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι μόνο εκεί για να εξυπηρετήσει την κυβέρνηση, είναι εκεί για να εξυπηρετήσει ε, τον λαό του Ιράκ. Πολλές από τις δραστηριότητες μας λοιπόν περνούν στους απαλούς τομείς όπως η δημιουργία θεσμών, το εκλογικό σύστημα, η προστασία των μειονοτήτων, ιδιαίτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά δεν είναι πολύ θεματικά. Κάποιες φορές στις συζητήσεις μας εστιάζουμε πολύ στην MEK και ή στην Ashraf, αλλά ωστόσο είμαστε ευγνώμονε για οποιαδήποτε στήριξη μπορεί να έχουμε για αυτά τα θέματα, όπω η δημιουργία των θεσμών, η πρόθεση των εκκρεμών ζητημάτων του συντάγματος, ο σχηματισμό του δεύτερου σώματος, του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της χώρας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εκλογικά σώματα. Όλα αυτά πολύ δύσκολα θέματα, τα οποία όμως δεν είναι θεματικά όπου εμείς έχουμε ένα γραφείο μέσα στο Συμβούλιο Εκπροσώπων, ε, το, στο Κοινοβούλιο μάλλον του Ιράκ, έχουμε γραφείο στο ανεξά, στην Ανεξάρτητη Επιτροπή ε, Εκλογών. προσπαθούμε να συμβουλέψουμε για την εκλογή των νέων επιτρόπων. Είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ερχόμαστε σε επαφή με τα μισμιονότητες της χώρας, είτε είναι χριστιανοί είτε άλλοι που υποφέρουν από διώξεις. Και προσπαθούμε να προωθήσουμε την νομοθεσία περιμενωτήτων που πρέπει να γίνει μέσα στο πλαίσιο του συντάγματος. Αυτές είναι οι βασικές μας δραστηριότητε. και η ανθρωπιστική πτυχή που τη συζητάμε πάντοτε μαζί σας εδώ για το στρατόπεδο Ασράφ είναι πολύ σημαντικό, ναι, αλλά δεν είναι η κύρια μας δραστηριότητα. Τώρα, για το στρατόπεδο Ασράφ μπορεί να διαβάσατε ότι προχτές έγινε η τρίτη κίνηση των κατοίκων του Ασράφ στο στρατόπεδο Liberty. Όσοι, για όσους δεν παρακολουθούν καθημερινά την κατάσταση, να σας πω από τον Απρίλιο και του 2011 τι έγινε επίθεση της Ιρακινής κυβέρνησης ε, στο Ασράφ με 40 νεκρούς και πολλές εκατοντάδες τραυματίες. Η κυβέρνηση τότε αποφάσισε να εκενώσει αυτό το στρατόπεδο μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου και γι' αυτό εμείς ε, δραστηριοποιηθήκαμε, μας ζήτησαν να δράσουμε και να προλάβουμε ένα τέτοιο άλλο γεγονός, όπως τον Απρίλιο. Τώρα, τα συμφέροντα είναι πολλά από όλες τις πλευρές. Η κυβέρνηση του Ιράκ τι θέλει. Το MEK να βγει εκτός του επικράτειας του Ιράκ, να φύγει από την χώρα και να κλείσει το στρατόπεδο Ασράφ. αυτή η εξεδαφικότητα ε, θεωρούν ότι θα πάψει την βία, θα σταματήσει τη βία. Ε, εμείς συνεργαστήκαμε με την κυβέρνηση και υπογράψθηκε ένα μνημόνιο συνεννόησης ε, στις 25 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους. Στόχος της κυβέρνησης είναι να γίνει μια κίνηση από το στρατόπεδο Άσραφ στο στρατόπεδο Liberty και να μείνει ένα από τα δύο στρατόπεδα. Γι' αυτό το σκοπό ο Πρωθυπουργό Μαλέκη επέκτανε, παρέτεινε την προθεσμία που αρχικά είχε ορίσει το για το Δεκέμβριο του 2011 στα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους. Και η προσπάθεια της μετακίνησης διέπεται από, δι... από μάλλον ε, συνίσταται σε τρία βήματα. Πρώτον, μετακίνηση και κλείσιμο του στρατοπέδου Ασράφ μέχρι τα τέλη του Απριλίου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και είμαστε σε αυτό το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να δώσει στην ε, ΥΠΑ του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες τη δυνατότητα να ε, εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης καθεστώτος ασύλου στους πρόσφυγες που το επιθυμούν και μετά από την ολοκλήρωση αυτής της, ε, της διαδικασίας να δοθεί δυνατότητα εγκατάστασης αυτούς τους πρόσφυγες σε άλλες χώρες εκτός Ιράκ. Αυτό είναι το μνημόνιο που έχει υπογραφεί. Τώρα, η κυβέρνηση του Ιράκ έχει δύο άλλες αρχές. Ε, πρώτον, κυριαρχία του κράτους του Ιράκ κατέστησαν σαφές ότι δεν θα ανεχθούν να υπάρξει ένα παραστατικό στρατόπεδο που δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση ή όπου θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση μόνο με τη βία, όπως τον Απρίλιο πέρυσι. Άλλη αρχή που επίσης νομίζω είναι κατανοητή για όλους, κάθε Ιρακινός πολίτης ή κάθε πολίτης που ζει στην επικράτεια του Ιράκ πρέπει να σέβεται τις Ιρακινένους νόμους, δηλαδή την αρχή της ε, κυριαρχίας και το εναρχείο ότι κάθε πολίτης πρέπει να υπακούει στους νόμους της χώρας. Τώρα είμαστε στη διαδικασία της ε, μετεγκατάστασης του ε, στρατοπέδου των, των, των Ασράφης στο Λίμπερτι. Εμείς τώρα παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία με τους επόπτες του ΟΗΕ, τόσο για τη μεταφορά όσο και για την κατάσταση στο στρατόπεδο ΑΣΡΑΦ. Έχουν καθημερινή έκθεση δίνεται για το τι γίνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας με την κατάσταση και, και τι βλέπουν εντός του στρατοπέδου, ποια είναι τα παράπονα φτάσαμε, καταφέραμε να φτιάξουμε μία δομή διαχείρισης ε, όπου αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα. Αυτή, έτσι γίνεται η παρακολούθηση. Αυτή είναι μία συνιστόσα. Η δεύτερη είναι ο καθορισμός ε, του καθεστώτος των προσφύγων όπου η ΥΠΑΤΗ για τους πρόσφυγες έχει διαφορετική τοποθεσία εκτός του στατοπέδου Λίμπερτη, ένα άλλο μέρος όπου μπορεί να πάρει συνεντεύξεις από τον κόσμο και τελικά μπορεί αυτό να οδηγήσει στην αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα. Και η τρίτη λειτουργία του ΟΗΕ και αυτό είναι ένα είδος ρόλου διευκόλυνσης. Έχουμε εδώ δύο αρχές. Για μας είναι μια υπόθεση ανθρωπιστική. Εμεί δεν ανακατευόμαστε στην πολιτική ω ΟΗΕ. Γνωρίζουμε φυσικά πως η κυβέρνηση του Ιράκ θεωρεί ότι οι όσοι διαμένουν στο στρατόπεδο Ασράφη θεωρούνται παράνομα διαμένονται στη χώρα και ταυτόχρονα την ε, PMOI δηλαδή τους Μονταχετίν ως τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό καθορίζει τις δράσεις τους, τις ενεργειές τους. Θεωρούν δηλαδή ότι όσοι διαμένουν εκεί είναι παράνομοι, αλλοδαποί στη χώρα και ότι η οργάνωση στην οποία ανήκουν είναι τρομοκρατική. Και γι' αυτό και εμείς από το ΝΟΙΕ δεν ανακατευόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Για μας πρόκειται για είναι 3.100-200 άνθρωποι, ανθρωπιστική κατάσταση, κρίση και, σε αυτήν, και, έτσι αν αντιδρούμε, όπως και για τους εκτοπισμένους, τους εσωτερικά εκτοπισμένους κτλ. Δεν ε, ανακατευόμαστε, όπως σας είπα, στην πολιτική πτυχή του θέματος. Και έπειτα, θα ήθελα επίσης να σας πω ότι υποστηρίζεται η εθελοντική μετακίνηση. Οι εναλλακτικέ δεν είναι πολύ καλές. Το να μείνει κανείς δηλαδή εκεί και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να μετακινηθεί αναγκαστικά κάπου αλλού, σε φυλακές ή αλλού. Ή ε, να επιλέξει αυτή την προσφορά του μνημονίου συνεννόησης και να μετακινηθεί από το στρατόπεδο Ασράφ σε κάποιο άλλο υπό ε, την προϋπόθεση πως η UNHCR θα τοποθετηθεί εκτός της χώρας. Η επανεγκατάσταση είναι το θέμα, το πρόβλημα, όχι τα μεμονωμένα προβλήματα που υπάρχουν βέβαια, δεν το αρνούμε, αλλά την επόμενη Παρασκευή στη Γενέβη έχουμε μια διάσκεψη των χωρών που παραδοσιακά ε, δέχονται πρόσφυγες. Και αυτό είναι και ο πυρήνας του προβλήματος τόσο η e και η κυβέρνηση, όσο και η κυβέρνηση του Ιράκ συμφωνούν πως η διαδικασία επανεγκατάστασης θα πρέπει να γίνει ε, και θα πρέπει αυτό να γίνει εκτός Ιράκ. Αυτή είναι η βασική μας δουλειά. Εμείς διευκολύνουμε, είναι μια οδυνηρή διαδικασία μετεγκατάστασης των ε, ε, συγκεντρωμένο στρατόπεδο Ασράφ στο στρατόπεδο Λίμπερτι και καταλαβαίνω πως όσοι ζουν εκεί και ζουν εκεί εδώ και 25 χρόνια και πρέπει να εγκαταλείψουν τις ρίζες που έχουν εκεί, δεν είναι πολύ εύκολο για να μετακινηθούν αλλού. Ωστόσο, είναι ένας τρόπος για ειρηνική επίλυση αυτού του, πολιτικού προβλήματος μέσω του στρατοπέδου Liberty προς το εξωτερικό. Τώρα βέβαια υπάρχουν προκλήσεις και υπάρχουν και ευκαιρίες όπως πάντοτε φυσικά. Πολλές επιστολές παίρνω από εσά και από εσά όσον αφορά τα προβλήματα υποδομών, το ότι δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρισμού και οτιδήποτε άλλο. Εν μέρει όλα αυτά αληθεύουν, πολλά είναι υπερβολικά, αλλά εν μέρει αληθεύουν ότι οι Ιρακινοί πρέπει εδώ να ε, ενεργήσουν, να δράσουν και τους το θυμίζουμε. Και έπειτα θα πρέπει να υπάρξει και μια συνεργασία από πλευράς των κατοίκων του Άσραφ, αν συμφωνούν ε, σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να σας πω ότι οι ρακινές δυνάμεις, είτε είναι η αστυνομία είτε είναι στρατός, είναι πολύ υπομονετικοί κατά τη διάρκεια αυτή τη ε, οδυνηρή διαδικασία με την κατάσταση από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Παίρνει πάρα πολύ χρόνο, διότι η ασφάλεια είναι στα χέρια των Ιρακινών. Πρέπει να ελέγξουν όλα του τα προσωπικά αντικείμενα μέχρι ότου να φορτωθούν στα φορτηγά και στα λεωφορεία. Και πολλές φορές 70-80 οχήματα ε, ασθενοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία μετακινούνται σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Οι Ιρακινοί απασχολούν περίπου 9.000 εκεί και η υπομονή είναι πολύ απαραίτητη. Προσωπικά εγώ συμμετέχω αν υπάρχουν προβλήματα και συνοδεύουμε αυτή τη δικασία και δημιουργούνται προβλήματα κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης και την παρακολουθούμε πολύ στενά και πραγματικά προσπαθούμε να διευκολύνουμε την ε, ταχεία μετεγκατάσταση. Επίσης, για τον, την πλευρά του ΟΙΕ έχουμε προκλήσεις. Η διαδικασία της αρμοστίας για τους πρόσφυγες είναι πολύ αργή, εξακολουθεί να είναι πολύ αργή. Οι συνεντεύξεις παίρνουν πάρα πολύ χρόνο γιατί είναι πολύ περίπλοκο τα θέματα, αλλά αυτό ισχύει παγκοσμίω. Δηλαδή είναι στάνταρ που ισχύουν παγκοσμίω. Και η δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και θέλω αυτό να το τονίσω άλλη μια φορά είναι η διαδικασία επανεγκατάσταση είναι το τρίτο βήμα. Γιατί όταν αυτός ο κόσμος θα πάει στο στρατόπεδο Λίμπερτ, που δεν είναι τόσο καλό όπως ήταν το στρατόπεδο Άσραφ, θα πρέπει να φύγουν και από τη χώρα. Και κάνω έκκληση στα κράτη-μέλη, ώστε πραγματικά να ανοίξουν τα σύνορά τους και να τους δεχτούν ως πρόσφυγες. Η Μουτζαχεντίν του Ιράν διαπραγματεύονται τις μελλοντικέ κινήσεις και σε εκείνους κάνω έκκληση για να δείξουν την απαραίτητη διάθεση της συνεργασίας όσον αφορά την τοποθεσία, της υποδομές στο στρατόπεδο. Εμείς διαπραγματευθήκαμε για πολύ καιρό την παρουσία της αστυνομίας στο στρατόπεδο, τώρα έχει ρυθμιστεί. Οι συναντήσεις της διεύθυνση του στρατοπέδου ε, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματα και το πλεονέκτημα της διαδικασίας αυτής είναι ότι έχει δραστηριοποιηθεί το UNHCR, η υπηρεσία προς, η προσφύγων, έχουμε και έχει ενεργοποιηθεί, παρακολουθεί τα πάντα. Εμείς είμαστε εκεί παρόντες, με παρατηρητές και επόπτες και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί, δεν είναι μόνο ο ΙΕ, αλλά και οι πρεσβείς που απέχουν μόλις 30 λεπτά από το στρατόπεδο Ασράφ ε, στη Βαγδάτη και οποτεδήποτε προκύψουν προβλήματα ενημερώνονται, προειδοποιούνται και είμαστε σε στενή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κόμπλερ. Αναφέρατε μια πρώην συναδελφό μας εδώ πέρα, ε, την οποία τηλεφωνήθηκα πριν από δύο ημέρες και θέλω να σας πω πως δεν παραπονιέται, αλλά όταν βλέπω τις συνθήκες εκεί πέρα των εκπροσώπων της Ένωσης 6 ε, άτομα σε, σε ένα κουτί στο εσωτερικό της, στην αυλή της Βρετανικής Πρεσβείας. Ε, δεν νομίζω πως είναι οι συνθήκες αυτές. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε και με τους υπεύθυνου της εξωτερικής υπηρεσία. Είναι εξαιρετικό το ότι αυτή η γυναίκα ε, κάνει αυτή τη δουλειά υπό αυτές τις συνθήκες. Είναι αξιοθαύμαστο. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να, το, να το πούμε. Το λόγο έχει τώρα κ. Στίβενσον, επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, με Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Να καλωσορίσω και εγώ και τον κύριο Μάρτιν Κομπλερ και τον κύριο Νταν Φρίντ για το ότι ήρθαν από πολύ μακριά για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση στο Ιράκ και στο στρατόπεδο Άστραφ. Συναντήθηκα χτες με δύο ανθρώπους από το γραφείο του Πρωθυπουργού Νούρι Αλμαλίκη. Και μιλήσαμε για την κατάσταση που φαίνεται πως επιδεινώνεται από τοπική εξέγερση. Αυξάνεται. Όταν ήμουν πέρσι στη Βαγδάτη με τον Μάριο Μαουρό και τον Γιάλκο Κατσίν και τον Τζον Μονταλτό μας είπαν τότε πως οι Αμερικανοί θα έφυγαν τέσσερις ώρες τη μέρα είχαν ρεύμα στη Βαγδάτη, νερό πόσιμο δεν υπήρχε πουθενά στη χώρα. Εκπαίδευση δεν υπήρχε, οι υποδομές κατέρεαν. Η χώρα και ήταν σε κακή κατάσταση. και μου είπαν πως η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί παρά το ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο αυξάνονται αλματοδός. Αλλά διεθνώς το Ιράκ είναι η δεύτερη πιο διεφθαρμένη χώρα στον πλανήτη μετά τη Σομαλία. Και πρέπει να ρωτιέται κανείς που πάνε αυτά τα λεφτά. Είναι κρίμα το ότι δεν υπάρχει χρηστή διοίκηση στη χώρα και από ό,τι φαίνεται έχουμε συγκρούσει μεταξύ φατριών. Θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπατε κύριε Πρόεδρε. Η Γιάννα Ιμπάσκοβα, η πρώην συνάδελφός μας, κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά υπό συνθήκες φρικτές σε ένα νοικιασμένο γραφείο στη Βρετανική Πρεσβεία που κανείς από εμά δεν θα πήγαινε να δουλέψει, σας διαβεβαιώ. Με έξι μόνο συναδέλφους ακούσαμε πριν την, τα της παρουσίας ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης στα Μπαρμπέντος, όπου υπάρχουν δεκάδες διπλωμάτες. Ε, δεν είναι κατάσταση αυτή. Συμφωνώ πλήρω με αυτά τα οποία είπε ο Μάρτιν Κόμπλερ. Πρέπει να στείλουμε περισσότερους ανθρώπους εκεί και να ανοίξει γραφείο και στο Κουρδιστάν, στα Μαρμπίλ. Να στραφούμε τώρα στο θέμα του ΑΣΡΑΦ γιατί είμαι και σε επαφή με την Πατρίσια Λόμπαρτ από την Κομισιόν και ευχαριστώ και τον Μάρτι Κόμπλερ για τις συχνές μας επαφές, αλλά εμένα με ενημερώνουν και από το στρατόπεδο Άσραφ και για τους 1190 ε, που έχουμε μετακομίσει στο στρατόπεδο Liberty η κατάσταση της ε, τελευταίας μετακόμισης που αφορούσε 400 άτομα. Τους είπαν πως έπρεπε να μετακομίσουν την παραμονή του Νευρός μεγάλη γιορτή για τους Ιρανούς, αλλά παρόλα αυτά ήθελαν να συνεργαστούν και συμφώνησαν. Αλλά όπως είπε και ο Μάρτιν Κόμπλερ, η μεταφορά αυτή χρειάζεται μέχρι και 50 ώρες όταν ερευνήσουν όλα τους τα προσωπικά αντικείμενα, τα δακτυλικά αποτυπώματα κτλ. Όταν φτάσουν στο στρατόπεδο Liberty μετά από δύο ώρες και περισσότερο ίσως, τους άφησαν να κάθονται στο λεωφορείο άλλες 6 ώρες, δεν τους άφησαν να κατέβουν να πάνε στην τουαλέτα καν. Το αποτέλεσμα ήταν πως χτες ένας από τους Ιρανούς, ο κύριος Μουσταφιάν, πέθανε από καρδιακή προσβολή στα 45 του. ο γιατρός είπε πως αυτό ήταν λόγω της κούρασης και του άγχους ε, λόγω όλης αυτής της διαδικασίας και θεωρώ πως όλα αυτά είναι λυπηρά. Πολλοί άνθρωποι μου λένε μα γιατί η Ιρακινή κυβέρνηση όταν ήθελε να ξεκαθαρίσει το, το Άστραφ και να βγάλουν την οργάνωση αυτή εκτός του Ιράκ γιατί δεν τους ανέκριναν στο Άστραφ γιατί όλες αυτές οι βλακίες να μετακομίζουν από εδώ και από εκεί σε αυτή τη μικρή εγκατάσταση μισού τετραγωνικού χιλιόμετρου γιατί οι υποδομές αυτές δεν κάνουν δεν επαρκούν ούτε καν για τους 1.200 που είναι εκεί τώρα, πόσο μάλλον τους 3.300 που θα προσθεθούν. Μα είχαν πει πως θα ήταν ε, εκεί πέρα ένα μετεβατικό στρατόπεδο για λίγους μήνες και τώρα μας λένε πως όπως ανακρίνει και παίρνει συνεντεύξεις η ύπατη αρμοστία για να αποφασίσει ποιος είναι πρόσφυγας ε, μιλάνε με έναν άνθρωπο τη μέρα. Δηλαδή με αυτό το ρυθμό 3.300 άτομα θα χρειαστούν 8 χρόνια. Δεν επαρκεί αυτό για να ζει ο κόσμος 8 χρόνια, ούτε 8 μήνες. Και πρόκειται για παραβίαση του μνημονίου μεταξύ του ΟΗΕ και της κυβέρνησης του Ιράκ. Και έχει παραβιαστεί και άλλες φορές, γιατί μας είπαν πως οι άνθρωποι αυτοί θα είχαν ε, ε, τα αγαθά τους όποιος, οποιοδήποτε ε, πολίτης ε, του Ιράκ, δεν τους δίνουν οικοδομικά υλικά, λέγαν πως θα φρόντισαν μόνοι τους την υποδομή, αλλά δεν μπορούν να έχουν εργαλεία, ούτε οικοδομικά υλικά, Οπότε η υποδομή δεν μπορεί να βελτιωθεί. Και οι παρατηρητές του ΟΗΕ Εντάξει, καλό να έχουμε παρατηρητέ του ΟΗΕ, αλλά όταν στέλνουν τι ε, αναφορέ του στην κυβέρνηση του Ιράκ δεν συμβαίνει τίποτα. Εμένα μου έστειλαν την προηγούμενη εβδομάδα μία λίστα με 59 καταγγελίε, χωρί καμία αντίδραση από την κυβέρνηση του Ιράκ. Έχουμε τώρα ε, έτοιμα από τους 800 αρχικούς ε, κρατούμενους στο στρατόπεδο Λίμπερτι που υπέγραψαν και λένε μην επιτρέψετε σε άλλους να έρθουν εδώ πέρα μέχρι να έχουμε κάποια αξιοπρέπεια στις υποδομές. Να έχουμε νερό, αποχέτευση και οικοδομικά υλικά. Ειδικά εάν είναι να εξαναγκαστούν να ζήσουν εκεί πέρα για μεγάλες περιόδους. Τέλος, να πω κύριε Πρόεδρε το εξή. Αντιλαμβάνομαι πλήρως πως υπάρχουν πρωινές συναντήσεις κάθε μέρα με τις καταγγελίες αυτές στο στρατόπεδο Λίμπερτ. Οι πρωινέ συναντήσεις είναι υπό την προεδρία του συνταγματάρχη Σαντέκ, ηγέτη μίας από τις σφαγές του Ιουλίου του 2009 και Απριλίου του 2011, τις οποίες ανέφερε ο Μάρκ Κόμπλερ. Αυτός ο άνθρωπος διευθύνει τις πρωινέ συναντήσεις και αντιλαμβάνεστε, όταν ήταν επικεφαλής σφαγής, δεν ε, ασχολείται και με τις καταγγελίες αυτές τι οποίε απλά αγνοεί η κυβέρνηση του Ιράκ. Οπότε η κατάσταση δεν είναι σωστή, δεν μα τιμά και πρέπει να πω προ τον Μάρτιν Κομπλέρ, αντιλαμβάνομαι την ευθύνη σα, η οποία επεκτείνεται σε ολόκληρο το Ιράκ βεβαίω, και είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα χωρί να χρειαστεί να ασχοληθείτε και με το Άσραφ αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν τελείω από το Ιράκ και το εμπόδιο είναι η κυβέρνηση του Ιράκ η ίδια πρέπει να του ασκήσουμε πίεση. Ο ΙΕ δηλαδή, για να γίνουν πιο συνεργάσιμοι. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάουρο τώρα, ο εισηγητής μας, αλλά παρακαλώ, ε, έχουμε εξαντλήσει σχεδόν το χρόνο μας. Γι' αυτό σας να παρακαλώ, συνάδελφοι, μην ξεπεράσετε το δίλεπτο ο καθένας. Ο κύριος Μάουρο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μείνω στα δύο λεπτά. Ήθελα να κάνω ερωτήσεις στον Μάρτιν Κόμπλερ σε σχέση με τα όσα πιστεύω θα είναι τρεις συγκεκριμένες πτυχές που αφορούν τις αρμοδιότητες, το ΙΕΣ, το ιεροκοινό ε, πεδίο. Το πρώτη ερώτηση αφορά τον ίδιο τον ΟΗΕ. Ποια είναι η στρατηγική συμφιλίωση ανάμεσα σε Σουνίτες και Σιήτες που προτίθεται να προωθήσουν τα Ηνωμένα Έθνη δεδομένες της περιθωριοποίηση των Σουνιτών στην Ιρακινή κοινωνία που έχει ε, συνέπειες που διαρκούν ε, τρομοκρατία και ρήξη ε, στο Ιράκ, κυρίως σε μια πόλη όπως η Βαγδάτη. Και έπειτα, δεύτερη ερώτηση. Έχετε την εντύπωση ότι μπορεί να ξεσπάσει μια ανθρωπιστική κρίση, ότι δηλαδή λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στην Συρία μπορεί να υπάρξει μια ροή Ιρακινών που κατά χιλιάδες ζουν στη Συρία και θα θελήσουν να επιστρέψουν προς το Ιράκ βιαστικά, βιαστικά και με καταστροφικές συνέπειες. Και ε, ως προς αυτό τι σκοπεύετε να κάνετε. Τρίτη μου ερώτηση και δεν θέλω να δημιουργήσω διπλωματικά ζητήματα ανάμεσα στον ΟΗΕ και την ΕΕ. Όμως ειλικρινά η Ευρώπη πριν από πολλά χρόνια διχάστηκε για το Ιράκ. Ε, δηλαδή αντιμετωπίσαμε αυτή την κρίση διχασμένη με συνέπειες που δεν ήταν ε, θετικές. Αν υπάρχει μια, ένα μέρος όπου υπάρχει αίσθηση της κοινή εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Ιράκ. Μήπως δεν νομίζετε πως ε, οι δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ είναι μικρές σε σχέση με τις προσδοκίες. Δηλαδή δεν είναι ένα μέρος όπου θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντα Ευχαριστώ. Ε, το αμερικό, αμερικανικό ενδιαφέρον στα τόπεδα Άσραφ και Λιμπερτή έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ενδιαφέρονται και φροντίζουν για την ε, ασφαλή διαμετακόμιση των κατοίκων του στρατοπέδου Ασράφ στο Λιμπερτή και επίσης την, ε, την ασφαλή έξοδο των ανθρώπων αυτών και από, από το Liberty εκτός του Ιράκ. Και έχουμε είτε δημερώσει είτε πολυμερώς συζητήσεις με το Ιράκ, αλλά σε συντονισμό και υπό την αιγύδα των Ηνωμένων Εθνών. Επισκεφθήκαμε το στρατόπεδο, επισκεφτόμαστε τακτικά το στρατόπεδο Liberty και έχουμε γνώση της κατάστασης που επικρατεί. Οι συνθήκες στο στρατόπεδο Liberty επιδέχονται βελτιώσει φυσικά, αλλά δεν είναι τόσο κακέ όσο παρουσιάζονται μερικές φορές. Το κλειδί της επιτυχίας πάντως δεν είναι στην ανάλωση της ενέργειάς μας για τις συνθήκες στο στρατόπεδο Liberty ή στις πομπέ, στις ορδέ οχημάτων μεταξύ στρατοπέδου ΣΡΑΦ και Λίμπερτι. Νομίζω το κλειδί της επιτυχίας είναι η επανεγκατάσταση όσο περισσότερο ανθρώπων γίνεται στο στρατόπεδο Λιμπέρτη και μάλιστα το συντομότερο δυνατό μέσω της διαδικασίας της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ και φυσικά ασφαλή και σύντομη έξοδό τους και από το Ιράκ. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και όπως είπε ο κύριος Στίβενσον είναι χρονοβόρα, είναι πολύ αργή αλλά είναι σημαντικό οι κάτοικοι του στρατοπέδου Λίμπερτη να συνεργαστούν πλήρως με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ του λεχθέντος. Η διαδικασία αυτή δεν θα στεφτεί με επιτυχία παρά μόνο αν οι κυβερνήσει της Ευρώπης και των ΗΠΑ και άλλων ενδιαφερομένων χωρών αν δεν αναλάβουν και τις δικές τους ευθύνες και κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη διαδικασία επαναγκατάστασης υπό την αιγίδα της ΙΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την ΙΠΑ τη αρμοστία του ΟΗΕ ώστε να μην παραμείνει κόσμος στο στρατόπεδο Liberty για πάντα. Και θα παρακολουθήσουμε τις συζητήσεις της Παρασκευής στη Γενέβη για να δούμε πού βρισκόμαστε και να δώσουμε την όθηση για περαιτέρω πρόοδο. Ευχαριστώ κύριο Σμιγκαρέλη. Ευχαριστώ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις ανεπάρκειες και τις αδυναμίες της που επισημάνθηκαν συνεχίζει τη δεσμευσή της για να στηρίξει την διάρθρωση και του Ιράκ και την δημοκρατική του μετάβαση. Τεράστια τα εμπόδια, το περιβάλλον στις γειτονικές χώρες δεν είναι το πιο πρόσφορο και το κλίμα, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στη Βαγδάτη παρά τις, ε, τους δημοσιονομικούς μας περιορισμούς. Προσπαθούμε να έχουμε και στέρεη διμερή σχέση μέσω της ε, ε, Σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Ιράκ που θα λάβει χώρα τις επόμενες εβδομάδες. Η συμφωνία αυτή θα μας δώσει και τη νομική βάση που αυτή τη στιγμή μας λείπει για να έχουμε μια σταθερή και στέρεη σχέση με το Ιράκ. Αν υπογραφεί η συμφωνία αυτή θα καταφέρουμε να διοργανώνουμε τακτικές συνεδριάσεις σε ε, επίπεδο υπουργών, υψηλόβαθμων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων, οπότε θα δημιουργηθεί ένα θεσμικό αρχιτεκτόνημα στέρεο και θα το αξιοποιήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συναυθεί η συμφωνία αυτή το συντομότερο δυνατό. Εν τω μεταξύ εφαρμόζουμε το μνημόνιο που είχε υπογραφεί εδώ και μήνες από τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας Oettinger με τον Υπουργό Ενέργειας του Ιράκ. Αυτό το μνημόνιο για την ενέργεια θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε τη σχέση με το Ιράκ σε ένα πολλά υποσχόμενο τομέα τον ενεργειακό και για τις δύο πλευρές. Και ευελπιστούμε ότι η διάσκεψη κορυφή τη 29η Μαρτίου της, ε, του Αραβικού Συνδέσμου που θα γίνει στη Βαγδάτη τον επόμενο μήνα θα λάβει χώρα τελικά. Γιατί χάρη στη διάσκεψη αυτή τη κορυφή το Ιράκ θα ανακτήσει τον περιφερειακό και διεθνή ρόλο που είχε για πολλά χρόνια. Και έχουμε και ένα πρόγραμμα συνδρομή που είναι περιορισμένη σε εμβέλεια αλλά είναι φιλόδοξο από άποψη τεχνική συνδρομή και ε, προαγάγει, στόχο έχει την προαγωγή της ε, ε, χρηστής διακυβέρνησης και την ανασυγκρότηση του Ιρακινού κράτους σε τομείς κλειδιά. Επίσης, μεριμνούμε ιδιαίτερως για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Και δύο λόγια τελικά για το στρατόπεδο Ασράφ. Έχουμε συνεχείς επαφές με τους ευρωβουλευτές, ιδιαίτερα με τον κύριο Στίβενσον που ασχολείται με το θέμα αυτό. Είπε ότι εκπρόσωπος ε, θέτει το θέμα τακτικά στους υπουργούς εξωτερικών, ώστε η διαδικασία επανεγκατάστασης που γίνεται υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της αρμοστίας στο ΙΕ ε, να έρθει σε αίσιο πέρας. Και έχουμε και συνεχείς επαφές με τους Αμερικανούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζοντας τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα το εξαιρετικό έργο του Μάρτιν Κόμπλερ που διαδραματίζει σε πάρα πολύ αντίξωες συνθήκες. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κοιτάξτε, έχουμε 10-10 ομιλητές. Και, πρέπει... και έχουμε και άλλο θέμα στην μερίσια διάταξη. Οπότε, και αν είναι να τα βουλέψουμε, θα παρακαλέσω τους αδέλφους να μιλήσουν για ένα λεπτό και να κάνουν ερωτήσεις αντί να κάνουν δηλώσεις. Αλλιώς δεν θα κάνουμε τίποτα. Κύριε... Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε πραγματικά ότι για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα ε, θα αφιερώσουμε μόνο 10 λεπτά. Καλύτερα να το αναβάλουμε τελείως. Δεν έχει νόημα τόση λίγη ώρα για τόσο σημαντικό θέμα. We'll see. I think, you know, that we, if, if we... Βλέποντας και κάνοντας πάντως, αν ε, Σεβαστείτε το χρόνο. Τι να σας πω, εγώ έλαβα την Προεδρία στη μέση της συζήτησης περίπου. Κάνω ό,τι μπορώ, τι να κάνω. Δεν είναι προσωπική μορφή, κύριε Πρόεδρε. Αλλά όχι βλέποντας και κάνοντας, Σας αποφασίσουμε. Δεν είναι δικό σας λάθος, φταίξιμο. Παρακαλώ ένα λεπτό και να θέσετε ερωτήσεις. Ο κύριος Αλαφράνκα, ευχαριστώ εντάχει. Σημείωσα ε, τις παρατηρήσεις για το γενικό πλαίσιο των σχέσεων, τις προσπάθειες του ΟΗΕ, τη συμφωνία σύνδεσης που θα υπογράψουμε με το Ιράκ, τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης αυτής. Θα ήθελα να αναφερθώ στην κατάσταση στρατόπεδο, στα στρατόπεδα Ασράφ και Λίμπερτι. Καλό είναι να σημειώνουμε αυτά που ακούμε και να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες, αλλά θα πρέπει να, να αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες δράσεις ε, που θα αποτρέπουν ε, τέτοια θλιβερά περιστατικά όπως αυτά που μας περιέγραψε ο κύριος Στίβενσον. Έχουμε μια κατάσταση ανθρωπιστική. Δεν είναι θέμα μόνο οριοθέτηση αρμοδιοτήτων, ποιο είναι υπεύθυνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν θα πρέπει ο ένα να στέλνει τον μπαλάκι στον άλλον. Θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις για να ξεπεράσουμε μια κατάσταση. Είχαμε σφαγή και οι συνθήκες, οι ε, ανθρωπιστικές συνθήκες αυτών των ανθρώπων είναι πραγματικά επισφαλέστατες. Παρακαλώ κύριε Κόμπλερ, Κάντε ό,τι μπορείτε ώστε σε συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ πρόσωπο να λυθεί αυτό το πρόβλημα με την καλή βούληση και με την κινητοποίηση των απαραίτητων μέσων και πόρων για να βρεθεί μια λογική και δίκαιη λύση που θα λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα που έχουν αυτοί την άνθρωποι ως πρόσφυγες. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Για ένα λεπτό. θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέσβη για την εισαγωγή που έκανε για ολόκληρη αυτή την εικόνα στο Ιράκ και εγώ ως συγγήτρια αυτού του κοινοβουλίου το 2008 είχα κάνει μια έκθεση με συντριπτική πλειοψηφία για το ρόλο της Ένωσης στο Ιράκ. Και συμφωνώ πλήρως μαζί σας και θα έλεγα πώς πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή να αναπτύξουμε τη σχέση με το Ιράκ που βεβαίως απαιτεί τόσο μεγάλη προσοχή. Και συνεχώς ασχολούμαστε με ένα ζήτημα, όσο σημαντικό και αν είναι. Εντάξει, είναι σημαντικό, το αναγνωρίζω. Ε, το να εγκατασταθούν κάπου αλλού αυτοί οι άνθρωποι από το στρατόπεδο Άστρεφ. Γιατί ως συγκήτρια θεωρώ πως είναι πολύ ευαίσθητο το ζήτημα για το Ιράκ και τη σχέση με το Ιράν και για τους ίδιους του Ιρακινούς γιατί δεν ε, ασχολούμαστε με φυσιολογικούς πρόσφυγες, να το ξέρουμε αυτό. Μιλάμε για πολύ φανατικούς ανθρώπους, που βεβαίως πρέπει να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, αλλά πρέπει να τα γνωρίσουμε πως έχουν πολύ φανατική προσέγγιση. Δεν επιτρέπουν, παραδείγματος χάρη στους συγγενείς, να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους. Ελπίζω να αφιερώσουμε την ενέργειά μας να εστιάσουμε σε αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Πρέσβης. Να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας να επιτρέψουν τη μετεκατάσταση αυτών των ανθρώπων γιατί χωρίς αυτό δεν θα λύσουμε το πρόβλημα του στρατοπέδου Άστραφ αν είναι Λίμπερτη. Σας ευχαριστώ κυρία Λοχμπίλερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για ένα λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας κύριε Κόμπλερ δύο ερωτήματα. Το ένα αφορά τα πολλά άλλη τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ποιο βαθμό υπάρχουν ανεξάρτητα όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πώς έχει κατάσταση στις φυλακές. Όλο για βασανιστήρια ακούμε. Και για το Άσραφ. Υπάρχουν προσφορές από συγκεκριμένα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι με τους κρατωμένους στο στρατόπεδο Άστραφ ή ε, Λίμπερτι. Ευχαριστώ κύριε Λαντσμπέργκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατευθείαν σε ερωτήσεις θα περάσω. Τι ενδιαφέρον έδειξε η λιμπερτη ευχαριστω κυριε λαντσμπεργκης ευχαριστω κυριε προεδρε κατευθειαν σε ερωτησεις θα περασω τι ενδιαφερον εδειξε η κυβερνηση του Ιράκ, ε, υποτίθεται κυβέρνηση κυρίαρχου κράτους ε, και όχι δορυφόρου του Ιράν, να κλείσει και να καταστρέψει το στρατόπεδο Άσραφ. Δεν θα μπορούσαν ε, οι Ιρανοί να έχουν καθεστώς πρόσφυγα και να συνεχίσουν να ζουν στο Ασράφ και από εκεί να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες. Και ποια η διαφορά μεταξύ της τωρινής κατάστασης των 1200 Ιρανών που εκδιώχθηκαν από το Άσραφ στην μικρή βάση Λίμπερτη σε σύγκριση με μια φυλακή με εχθρικούς φύλακες και υπάρχει κάποια ιδέα να αλλάξει το όνομα της φυλακής από Λίμπερτη σε κάνα πιο κατάλληλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγκίνης και ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα από τα προβλήματα και θα συμφωνήσετε κύριε Κόμπλερ είναι πως ε, αναγνωρίζονται ακόμα από τις ΙΠΑ και το Ιράκ ε, ως ε, τρομοκρατική οργάνωση και έτσι έγιναν οι σφαγές του 2009 και του 2011. Να ρωτήσω τι εγγυήσεις έχετε πως όταν μεταφερθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουμε επανάληψη των γεγονότων του 2009 και του 2011. Εμείς μπορεί να χαιρόμαστε για τη μετακόμιση, αλλά ο φόβος είναι πως μόλις γίνει μετακόμιση θα υπάρξει άλλη μία επίθεση. Και τέλος, συμφωνείτε πως όταν συναντηθήκατε με εμένα και άλλους τρεις συναδέλφους πως υπήρχε μία εγγύηση για ηλεκτρισμό, αποχέτευση και ίδρυυση πριν ε, λάβει η χώρα η μεταφορά και δεν ισχύει αυτό. Χρειαζόμαστε μια εγγύηση πως αυτό θα συμβεί σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ. Τα γεγονότα της Τρίτης, τα χθεσινά δηλαδή, για τα γεγονότα αυτά, τους 50 νεκρούς δηλαδή, ανέλαβε την εθνική Αλκάιντα. Ζητώ συγγνώμη για την αδαιμοσύνη μου, αλλά στο αγώνα κατά της Αλκάιντα με τη βοήθεια των μυστικών υπηρεσιών. Πώς γίνεται ο συντονισμό υπεύθυνο για τον αγώνα αυτό, σε ποιο στηρίζεται η, Ιρανική, η κυβέρνηση. Η Γιουνάμι, ο ΙΕ, έχει κάποιο ρόλο εκεί. Η ΙΠΑ, ποιος βοηθάει το Ιράκ στον αγώνα κατά της Αλκάιντα. Είναι πολύ ανησυχητική αυτή η κατάσταση. Γιατί το Ιράκ έχει σύνορα με τη Συρία και όταν βλέπουμε τα γεγονότα της Συρίας δεν μπορούμε παρά να ανησυχούμε σε ό,τι αφορά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Θα μπορούσατε να διαφωτίσετε κάπως για το θέμα αυτό. Thank you very much. Ε, please. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση για τη θανατική ποινή. Το Ιράκ είναι μία από τις χώρες με τις περισσότερες καταδίκες σε θανατική ποινή. Έχω τα νούμερα της Διεθνούς Αμνηστίας. Πάνω από 300 άτομα καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν τα τελευταία 6 χρόνια. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η πολιτική του ΟΗΕ σε σχέση με αυτό στο Ιράκ και τι σκοπεύετε να κάνετε για να πείστε τους Ιρακινούς για την αναγκαιότητα της κύρωσης ε, του καθεστώτος του Διεθνούς ε, Ποινικού Δικαστηρίου. Είχαν πει το 2007 θα το κάνουν, αλλά ακόμα τίποτα. Και κάτι ακόμα για την βία μεταξύ των φίλων. Τεράστιο πρόβλημα. Εγκλήματα τιμής ε, και τα λοιπά. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως οι αρχές του Ιράκ θα αναλάβουν δράση σε αυτό το μέτωπο και κύριε Πρόεδρε κάτι για τις μειονότητες ε, είπατε πως υποφέρουν μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος σας ε, ευχαριστώ κύριε Κέλλαμ. ευχαριστώ να πω πόσο εκτιμώ τις προσπάθειές σας κύριοι Κόμπλερ και Φρίντ αλλά τώρα η κατάσταση πιέζει. Και έχει δημιουργηθεί τεχνητά γιατί υπάρχει ένας μήνας για τη μεταφορά των ανθρώπων και έχουν γίνει συνεντεύξεις με λιγότερο από 100 από αυτούς και υπάρχει και η πίεση του Ιράν μιας τρομοκρατικής δικτατορίας θέλει να ξεφορτωθεί αυτούς τους ανθρώπους που είναι κατά του καθεστώτος. Αλλά το ερώτημα μου είναι, έχουν πρόσβαση σε δικηγόρους και γιατρούς, γιατί μόνο το χρειάζονται. Και βεβαίω προστηρίζω πλήρως την έκκληση όλων των συμμετεχόντων για να ανοίξουν τα κράτη-μέλη τα σύνορά τους και να δεχτούν αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Πέτερλε. Ε, ευχαριστώ. Περισσότερες από τις που ήθελα να κάνω έχουν ήδη γίνει. Και αναρωτιέμαι κι εγώ. Δεν ήταν δυνατόν να προετοιμάσουμε ένα κατάλογο από πριν να γίνει αυτό στο προηγούμενο στρατόπεδο. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν τόσο καιρό να μην έχει ετοιμαστεί ένας κατάλογος. Ε, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την τελική λύση του ζητήματος, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία πως μπορούμε να πούμε κάτι για την διασφάλιση ανθρωπιστικών συνθήκων. Είναι προφανές πως η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Ναι, αν βασιστούμε στις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Ελπίζω το ζήτημα αυτό να επιληθεί και με την προσεχή συνάντηση στην Γενέβη. Για εμά, τους ευρωβουλευτέ, είναι απογοήτευση αυτό. Εδώ και τόσα χρόνια συζητάμε τα ίδια πράγματα. Ελπίζουμε λοιπόν να σημειωθεί κάποια πρόοδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Κόμπλερ για τις πληροφορίες. Θεωρώ πως οι άνθρωποι που ζουν στο στρατόπεδο Άστραφ ή Λίμπερτι τώρα ε, αξίζουν αξιοπρεπή μεταχείριση, όποιο καθίστος και αν έχουν. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Υποστηρίζω πλήρως αυτό το οποίο είπε ο κύριος Στίβενσον για το ότι μετα πρέπει να ληφθούν, πρέπει να αποφύγουμε περαιτέρω περιπλοκές ε, στην κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Δεν έχω ερώτηση. Απλά δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας ε, του κυρίου Κόβλερ για να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σαλαφράγκα. Γνωρίζουμε πως έχετε πολλές δραστηριότητες έχετε λίγες ε, δυνατότητες όσον αφορά το στρατόπεδο Άσραφ, αλλά χρησιμοποιήστε το στο έπακρο για να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μετά τα όσα είπατε δεν έχουμε κάποια διαβεβαίωση πως θα γίνει κάτι για να αλλάξει η κατάσταση προς το καλύτερο. Ευχαριστώ κύριε Φαντάλαν. Νομίζω πως συμφωνούμε όλοι πως πρέπει να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση. Ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Κόμπλερ τι μπορεί να γίνει συγκεκριμένα. Δεύτερον, οι Ολλανδοί ευρωβουλευτέ ζήτησαν επισήμω από τον Υπουργό Εξωτερικών μα να προσκαλέσει ε, πρόσφυγες από το Ιράν και το Ιράκ να έρθουν στην Ολλανδία. Ελπίζω να κάνουν το ίδιο και οι άλλοι ε, συναδελφοί μας. Πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κόμπλερ, έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ λακωνικός. Θα ξεκινήσω με τα θέματα που δεν αφορούν το στρατόπεδο Άσραφ. Ο κύριος Μάουρο είπε τι, κάνει, τι κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη, η Γιουνάμι για την επανασυμφιλίωση, για την πολιτική διαδικασία της επανασυμφιλίωσης. Οι Σουνίτες αισθάνονται παραγωνισμένοι. Έχουμε τρία επιχειρήματα που τα αναφέρουμε μονίμως συνομιλητές μας. Πρώτον, θέλουμε μια διαδικασία που δεν θα αποκλείει κανέναν. Θα εντάσσονται σε αυτή οι Κούρδοι, οι Σουνίτες και οι Σύντες. Δεν θέλουμε ε, να παραγωνίσουμε κανέναν. Κανένας δεν θα πρέπει να παραμεριστεί. Φυσικά οι Σύντες είναι εξορισμού μέσα, ούτε οι Σουνίτες ούτε οι Κούρδοι. Το boycott που έχει κάνει η ομάδα Ιρακία στο, στο Ιρακινό Κοινοβούλιο και στην Ιρακινή Κυβέρνηση δεν ήταν καλή ιδέα γιατί όποιος βγαίνει θα πρέπει να ξαναέρθει, να ξαναμπεί. Και δεν ξέρω αν γίνεται πάντα σε καλύτερες συνθήκες αυτή η επιστροφή. Τελικά το βοηκοτάρισμα σταμάτησε. Υπάρχει και ζήτημα διαφάνειας. Όποιες και να είναι εξελίξεις θα πρέπει να είναι διαφανείς. Αν οι Κούρδοι, οι Σιήτες και οι Σουνίτες ε, καθίσουν, συζητήσουν και συμφωνήσουν για έναν οδικό χάρτη, θα πρέπει να δημοσιευτεί αυτός να μην αποκλείται κανένας. Όχι μποϊκότ και διαφάνεια. Αυτά είναι τα τρία ε, ζητούμενα που τα επαναλαμβάνουμε μονίμως στις συζητήσεις. Σε ό,τι αφορά το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Το Σύνταγμα προβλέπει σαφώς ότι θα πρέπει να υπάρχει και δεύτερη βουλή, δεύτερο σώμα στο Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει όμως τέτοιο δεύτερο σώμα στη Βουλή. Δεν έχει ε, εγκριθεί ακόμη το νομοσχέδιο για το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και ο ΙΕ ε, επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο θέμα της δεύτερης βουλής, γιατί η τάση της ε, σουνητικής συνιστώσας είναι να αποσχιστεί και να ε, κηρύξει ε, ή να, διεκδικήσει για τις περιφέρειες παρόμοιο καθεστώς με αυτό στις, στη Bundestag. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Όταν θα έχουμε και μια δεύτερη βουλή όπου οι κυβερνήτες τοπικοί θα έχουν το λόγο στην δεύτερη αυτή βουλή, θα χαλαρώσει κάπως η πίεση για την περιφερειοποίηση. Και αυτό το λέμε σε όλους τους συνομιλητές και ενδιαφερόμενους και το ε, διακηρύσουμε και δημοσίως. Κάτι που μας φέρνει μερικές φορές και σε δύσκολη θέση, αλλά ε, έχουμε το θάρρος της γνώμης μας. Άλλο θέμα, η ανθρωπιστική κρίση στη Συρία. Τη στιγμή αυτή δεν υπάρχει ε, ροή, μεγάλη ροή, μαζική ροή προσφύγων προς το Ιράκ. Είχαμε 700 με 800 χιλιάδες Ιρακινούς πρόσφυγες που διαμένουν στη Συρία αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνουμε τάση επιστροφής τους στο Ιράκ. Είμαι και συντονιστή σχεδόν ε, των οργανισμών και προγραμμάτων ε, και της ΥΠΑ της Αρμόστιας. Και αυτό θέτω στους συναδέλφους ως ερώτημα. Τι γίνεται με τους ε, Σύριους Κούρδους στο Βορρά. Περιμένουμε μαζικές επιστροφές Πάντως από κοινού με το Υπουργείο με τα, μετεγκατάστασης και μετανάστευσης είμαστε ε, έτοιμοι, προετοιμαζόμαστε να δεχτούμε πρόσφυγες παρόλο που δεν υπάρχει τεράστια πλημμύριδα τέτοιων. Είναι περίπου 600 οι Σύριοι Κούρδοι που πέρασαν τα σύνορα στο Κουρδιστάν. Πρόσφατα επέστρεψε από εκεί, αλλά δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Δεν πρόκειται για κύμα μαζικής μετανάστευσης. Πάντως, ε, ε, Αποκινούμε κοινού με τις Ιρακινές αρχές ετοιμαζόμαστε ώστε αν υπάρξει μαζική διέλευση των συνόρων από πρόσφυγες να ε, τους υποδεχθούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ρώτησαν ε, η κυρία Λαχπίλερ και κάποιοι άλλοι. Ε, όταν διαπιστώνουμε καταστρατηγή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, διατρανώνουμε τη γνώμη μας. Το είπαμε και για την θανατική ποινή. Είπαμε, είπαμε προς την Ιρακινή κυβέρνηση θα πρέπει να καταργηθεί η θανατική ποινή και η πολιτική των, του ΟΗΕ είναι ένα μορατόριο για τη θανατική ποινή με σκοπό να βρεθεί μια λύση, να ισχύσει ένα νομικό καθεστώς που να απαγορεύει τη θανατική ποινή. Πάντως το πρώτο βήμα είναι ένα μορατόριο θανατικ, της θανατικής ποινής και αυτό το ε, δηλώσαμε και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό ε, εσωτερικών ε, και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρησιμοποιούμε και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να ε, διατρανώσουμε την αποτροπιασμό μας για την θανατική ποινή και μορατόριο στις εκτελέσεις, αμή τι άλλο. Τώρα, για την Επιτροπή υπάρχει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων στο, στην Ιρακινή Βουλή των Αντιπροσώπων και τώρα θα ε, επιλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επίτροπη της Ανεξάρτητης αυτής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είναι μια διαδικασία που έχει μεγάλη προβολή ε, και μάλιστα ε, οι δικοί μας εμπειρογνώμονες για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέχουν σύμβουλες και μίλησα με τον πρόεδρο της Ιρακινής Βουλής, τον κύριο Μουτζέιφη, παρόλο που μας πίεζε ο χρόνος και αποσαφηνίσαμε και οι δύο ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όχι μόνο για τη διεθνή κοινότητα που εκπροσωπώ εγώ, αλλά και για τι Ιρακινέ μη κυβερνητικέ οργανώσεις και για τον Ιρακινό λαό να οριστούν οι επίτροποι, τα μέλη δηλαδή τη της ανεξάρτητης Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συμμετέχουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων πάντω και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και αυτέ συμμετέχουν στην επιλογή με τον πιο διαφανή τρόπο όσο πιο διαφανή γίνεται τουλάχιστον, αυτό το ε, Συμβούλιο των Επιτρόπων της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί όπως θα φαντάζεστε. Πάντως επιμένουμε στην διαφανή διαδικασία, διαδικασία που θα χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, να είναι πραγματικά ανεξάρτητη αυτή η ανεξάρτητη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να έχει χρηστή οικονομική διαχείριση και ε, διαφανής ε, διαδικασία, ε, να έχει και μια διαφανή διαδικασία ελέγχου, εκλογής των επιτρόπων. Υπάρχει πρόβλημα με τις φυλακές, με τα βασανιστήρια, με τη διαφθορά. Δεν μιλάμε πάντα για βασανιστήρια, δεν είναι πάντα τα βασανιστήρια. Μερικές φορές καταβάλλονται χρήματα για να αποσπαστούν ομολογίες. Η διαφθορά είναι εκτεταμένη, το δηλώνουμε και δημοσίως ε, και θα υποβάλουμε και δημοσίως τις εκθέσεις ε, της UNAMI, του ΟΗΕ. Κατά πάσα πιθανότητα θα δυσαρεστήσουν πολλούς ε, οι εκθέσεις αυτές που θα δημοσιευθούν τον Απρίλιο για το Ιράκ από τη UNAMI. Το θέμα είναι ποιος ευθύνεται για τις επιδρομές αποκλειστικά και μόνο Ιρακινή, γιατί οι Αμερικανοί αποσύρθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου. Το θέμα της ασφάλειας αποτελεί πια αποκλειστική αρμοδιότητα των Ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας, του στρατού και της αστυνομίας. Και αν το συγκρίνουμε με μια κατάσταση πριν από τέσσερα χρόνια, το Δήμονο Γερμανό ε, πρέσβη στο Ιράκ, η κατάσταση σήμερα είναι πολύ καλύτερη, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πειθαρχία και η κατάσταση του Ιρακινού στρατού είναι πολύ καλύτερη από ό,τι πριν από μία τετραετία. Παρόλο που φυσικά μπορεί και να βελτιωθεί ακόμη. Βέβαια, κάθε τρομοκρατική επίθεση είναι μία επίθεση που καλό θα ήταν είχε αποφευθεί. Το είδαμε και χθε. 23 ε, Φεβρουαρίου είχαμε την προηγούμενη και χθε 20 Μαρτίου την άλλη. Ε, έχει μειωθεί κάπως συχνότητα των τρομοκρατικών επιθέσεων, αλλά παρόλα αυτά ε, υπάρχει βία. Όμως υπάρχει μια φθήνουσα κατάσταση και της βίας. Και επανέρχομαι στο στρατόπεδο Ασράφ. Δεν έγινε καμία δολοφονία στο στρατόπεδο Ασράφ. Δεν έγινε καμία δολοφονία. Όντως ε, κάποιος χθες το προέχασε τη ζωή του. Μετά την τρίτη κατάσταση. ένας κάτοικος του Ασράφ ε, πέθανε από καρδιακή προσβολή. Στις 8 Μαρτίου είχαμε επίσης ένα θάνατο στο στρατόπεδο Σραφ. Και υπάρχει ε, ιατρική περίθρεψη πολύ καλύτερη στο στρατόπεδο Λίμπερτι από ότι στο στρατόπεδο Σραφ. Υπάρχουν πολύ περισσότερα φάρμακα και καθημερινά ε, υπάρχει προσαγωγή σε νοσοκομεία εκτός του στρατοπέδου Liberty. Υπάρχει προσφορά ιατρικών υπηρεσιών δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειε για να μην μακρηγορήσω. Πάντω, το στρατόπεδο αυτό ε, είχε χωρητικότητα 5.500 ε, ε, και είχε ετοιμαστεί για 5.500 Αμερικανούς στρατιώτε, Ακόμη και προσωπικό του Γιουνάμι. Και μέχρι πέρυσι, στα τέλη του έτου και ηλεκτρισμό είχε και πόσιμο είδωρ και αποχέτευση. Νομίζω ότι από τη στιγμή που είχε υποδομέ για 5.500 ανθρώπου, έχει υποδομές και για 800. σε μία πρώτη φάση νομίζω ότι μπορεί να στεγάσει τα 800 άτομα που διαμέρουν εκεί. Τώρα, επειδή δεν είναι και πολύ συνεργάσιμη, κατ' εφημισμό το λέω, οι κάτοικοι ε, του στρατοπέδου ε, με τις ε, Ιρακινές αρχές, ε, δημιουργείται το πρόβλημα. Γιατί όταν υπάρχει μια διαρροή προσπαθούμε να τη διορθώσουμε, δεν αφήνουμε το πρόβλημα να οξυνθεί. Πάντως καθημερινά λαμβάνω αναφορές για το τι συμβαίνει εκεί. Εγώ δεν ανησυχώ ιδιαίτερω για την υποδομή, για τις υποδομές στο στρατόπεδο Λιμπερτή. Φυσικά κάποιες βελτιώσεις θα γίνουν, ιδιαίτερα στον ηλεκτρισμό. Θα πρέπει να δουλεύουν οι γεννήτριες, Γιατί θα αρχίσει σε λίγο η ε, θερμή περίοδος, ε, χρειάζεται κλιματισμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα προσωπικά αντικείμενα, η χρονοβόρα διαδικασία, κυρία Στίβενσον, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονό ότι οι κάτοικοι τη Άσραφ παίρνουν όλα του τα υπάρχοντα. Μπορεί και ένα άνθρωπο να έχει πέντε πνόσακου, για παράδειγμα. Και στην τελευταία μετεγκατάσταση είχαμε πρόβλημα γιατί έπαιρναν ακόμη και τι ε, λαμπτήρε του δρόμου, ακόμη και τι λιχνίε του, τα φανάρια πέραν μαζί του. Ε, βέβαια απαγορεύεται να έχουν πομπούς και δέκτες ε, φυσικά απαγορεύεται τα δομικά υλικά, αλλά μπορούν να έχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Και αυτό είναι όμω θέμα ερμηνεία και θέμα συνεργασίας μεταξύ των κατοίκων και των αρχών. Πάντω νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πιο ομαλά και πιο εύκολα αν ο καθένας είχε υπόψη του ότι ε, δικαιούται να μεταφέρει μόνο τα προσωπικά του αντικείμενα, τα προσωπικά του υπάρχοντα. Και επαναλαμβάνω, θα ήθελα να εξάρω την υπομονή των Ιρακινών αρχών και των Ιρακινών στρατιωτών. Θα πρέπει όμως ε, να υπάρχουν, να εφαρμόζονται οι κανόνες για τον περιορισμό ε, του τι μπορεί να μεταφέρει κανείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τις τραπεζαρίες, σίγουρα δεν είχαν και τις καταπληκτικές ε, τα καταπληκτικά εντευκτήρια και τραπεζαρίες ε, ε, του στρατοπέ, στο στρατόπεδο Λιμπερτή, αλλά οι κάτοικοι προφρόντισαν να... Ε, ενώ υπάρχει τέτοια τραπεζαρία που τη χρησιμοποιούσαν οι Αμερικανοί προηγουμένως και είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και προσφέρει όλα τα κομφόρ, οι επίτηδες, οι κάτοικοι του... Ε, οι πρώην κάτοικοι Ασράφιν, οι κάτοικοι του Λίμπερτι, προτίμησαν να μαγειρεύουν μόνοι τους έξω και επέμειναν να φέρουν και τους δικούς τους γιατρούς. Δεν θέλουν Ιρακινούς γιατρούς. Κάτι που φυσικά ε, δεν βρίσκει σύμφωνη την Ιρακινή κυβέρνηση γιατί οι δικοί τους ε, γιατροί μη Ιρακινοί δεν έχουν άδεια άσκηση επαγγέλματο. Και μας ρώτησαν γιατί δεν έγινε δυνατή αυτή η επιχείρηση της ΥΠΑ της Αρμοστίας στο ίδιο το στρατόπεδο ως ΡΑΦ. Και εγώ θέτω τις ερωτήσεις, αλλά η Ιρακινή κυβέρνηση όταν εγώ ανέλαβα τα καθήκοντά μου δεν αναγνώριζε καν την υπατή αρμοστία του ΙΕ. Όλοι οι κάτοικοι του Ασράφ υπέβαλαν τα ντοσιά για το, ε, για... το άσυλο, αλλά δεν αναγνωρίζονταν ως ετούντες άσυλο. Δεν αναγνωρίζονταν καν η ύπατη αρμοστία. Και εμείς ε, τα διαπραγματευτήκαμε. Στο στρατόπεδο Ασράφ δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσει η διαδικασία, γιατί έπρεπε να κλείσει το στρατόπεδο η διαδικασία της ΥΠΑ αρμοστής ήταν μόνο δυνατή εκτός του στρατοπέδου ΣΡΑΦ. Και άλλωστε οι κάτοικοι του, του στρατοπέδου Λίμπερτι αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες από την ΥΠΑ αρμοστή, αλλά όχι και από την κυβέρνηση του Ιράκ. Δεν έχουν τέτοιο χαρακτηρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το, τις φυλακές και τους εχθρικούς ε, δεσμοφύλακες. Όντως δεν υπάρχει ελευθερία διακίνηση στο στρατόπεδο και η κυβέρνηση του Ιράκ ε, θεωρεί τους κατοίκους ε, του Ασράφ ως, παράνο, ως παράνομους, Και όπως είπατε, θεωρούν την οργάνωσή τους, τους Μουζαχεντίν του Ιράν, ως τρομοκρατική οργάνωση και ρωτά τον ΟΗΕ τι κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες με κατοίκους ε, με αλλοδαπούς δηλαδή που είναι λαθρομετανάστες, ε, σε παρόμοια κατάσταση. Πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία τους λαθρομετανάστες. Ε, απαντήστε λοιπόν. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Λυπούμε που το λέω, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση για το ρεύμα για τον ηλεκτρισμό σε τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να επιβάλλουμε μια μετριοπάθεια, να παροτρύνουμε την κυβέρνηση να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, να εξασφαλίσει τις ε, υποδομές. Δεν υπάρχει καμία φυσικά εγγύηση ότι θα αποφευθεί νέα σφαγή. Πάντως θα θέλει την πολιτική μου κρίση, η Ιρακινή κυβέρνηση θέλει να φύγουν από τη χώρα οι κάτοικοι του στρατοπέδου Λίμπερτι. Και έχουν εκεί ε, παρατηρητές του ΟΗΕ, έχουν τον Γενικό πρόξερο, του ΙΠΑ πολύ κοντά, έχουν ε, πρεσβείες πολύ κοντά έχουν την Αμερικανική Πρεσβεία 2 χιλιόμετρα από το στρατόπεδο Liberty. Το δικό μας γραφείο βρίσκεται 30-40 λεπτά, όχι μία ώρα με το ελικόπτερο. Είναι υποστενή επιτήρηση οι Ιρακινές αρχές, οπότε αν δεν υπάρξουν προκλήσεις, η πιθανότητα να επαναληφθεί η σφαγή του Απριλίου είναι πολύ μικρή. Από τη στιγμή που υπάρχει διεθνής επιτήρηση, από τη στιγμή που και εσείς παρακολουθείτε με αμύωτο ενδιαφέρον την κατάσταση. Και α, αυτή τη που η Ιρακινή κυβέρνηση θέλει να ευοδοθεί η διαδικασία επανεγκατάσταση και ούτω ή άλλω πρέπει να κλείσει μέχρι τα τέλη Απριλίου το στρατόπεδο ΣΡΑΦ. Απευθύνω λοιπόν έκκληση προ όλου και τι κυβερνήσει, αλλά και του κατοίκου ε, των στρατοπέδων ΣΡΑΦ και Λίμπερτη να μην ε, λένε μόνο λόγια και να μην χρησιμοποιήσουν ρητορική γιατί δεν ε, θα λυθεί έτσι η κατάσταση. Καλή συνεργασία κανόνες που θα εφαρμόζονται, συνεργασία με τους παρατηρητές. Αντιλαμβάνομαι τις ευαισθησίες, γιατί υπάρχει δυσπιστία, υπάρχει δυσφορία και είναι λογική, είναι φυσιολογική αυτή η δυσπιστία, αλλά μόνο με καλή συνεργασία και καλή θέληση θα αποδοθεί η διαδικασία αυτή. Γι' αυτό και θα διευκολυθεί και το δικό μας έργο, γιατί αν μονίμως ε, ασκούνται επιθέσεις εις, βάρο, βάρος μας, αν έχουμε μια σελίδα στις New York Times εις βάρος ε, του ΟΗΕ ή μου προσωπικά ή του Ιράκ, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση. Θέλουμε ειρηνική λύση και όχι βίαιη λύση. Αυτό το ε, είπαμε και στους κατοίκους του Λίμπερτη, του Ασράφ και στην ε, Ιρακινή κυβέρνηση. Το Μνημόνιο Συνεννόησης μιλάει μόνο για ειρηνική λύση και όχι για βία λύση. Για να δω τις ε, σημειώσεις μου με ναι, πρόσβαση σε δικηγόρους. Δεν υπάρχει. Το έχω και εγώ και το φύγω με την κυβέρνηση του Ιράκ. Λένε πως δεν υπάρχει πρόσβαση σε δικηγόρους γιατί γιατί δεν υπάρχουν υποθέσεις. Κανείς δεν κατηγορείται για τίποτα. Οπότε αν υπάρξει κάποια διαδικασία βεβαίως θα έχουν και δικηγόρους. Αλλά δεν έχουν κατηγορηθεί για τίποτα. Κατά κατοικών... Δεν έχουν κατηγορηθεί για τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Οι ιατρικές υπηρεσίες, μεγάλο πρόβλημα. Ε, θα ρίνω. Mm. Τους ε, ενίκου εκεί πέρα να επιτρέψουν μια κλινική μέσα στο στρατόπεδο Liberty. Δεν επιτρέπουν οι ίδιοι ε, οι Ιρακινούς γιατρούς. Λένε εκτός του στρατοπέδου. Ε, δεν είναι δεκτό αυτό και από σκοπιά ανθρωπιστική. Και όσοι μιλάτε για ανθρώπινα δικαιώματα σας ενθαρρύνω να τους μιλήσετε να επιτρέψουν ιατρικές υπηρεσίες τόπου. Υπάρχουν δύο ασθενοφόρα, υπάρχουν δύο γιατροί, τέσσερις νοσοκόμες. Μεταφέρονται οι άνθρωποι στη Βαγδάτη και σε ειδικευμένους ιατρούς. Μπορούν να πάνε και σε ιδιωτική κλινική άμα θένε. αλλά εγώ πάντα λέω πως πρέπει να υπάρξει παροχή υπηρεσιών υγείας και δεν είναι σωστό να μην υπάρχει ε, κλινική εντός του στρατοπέδου. Βεβαίω λένε πως έχουμε τους δικούς μας γιατρούς, αλλά υπάρχει ένα σύστημα παραπομπής ε, στους γιατρούς, όπως σε οποιαδήποτε χώρα και εδώ πέρα. Δηλαδή πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι άσκηση, ε, άδεια άσκηση επαγγελματό. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν άδειες, έχουν άδειες στο Ιράκ. Η κυβέρνηση μας λέει εδώ μέσα είναι Ιράκ. Κυρίαρχη χώρα. Όλοι πρέπει να τηρούν τους νόμους. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ε, τελείωσε. Δύο σύντομε παρατηρήσει. Καταρχήν, οι πληροφορίε που έχει η κυβέρνησή μου συμφωνούν με τι πληροφορίε που μας έδωσε ο κύριος Κόμπλερ. Επίση, ε, δεύτερο θέμα, ε, αυτό έχει να κάνει με την, το καθεστώς της, ε, των οργάνωση Μουζαχετίν ε, υπό την Αμερικανική νομοθεσία. Ε, θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό το καθεστώς ε, είναι υπό αναθεώρηση. Την περασμένη χρονιά η, η Υπουργός Εξωτερικών Κλίντον έκανε την εξή δήλωση στο Κογκρέσο. Είπε ότι δεδομένων των συνεχιζόμενων προσπαθειών για μετακατάσταση των κατοίκων η συνεργασία των οργάνωσεων Μουζαχετίν είναι για την ειρηνική κατάσταση, θα είναι κλειδί, παράγοντας κλειδί σε σχέση με οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί σε σχέση με το καθεστώς της εν λόγω οργάνωσης. Θα ήθελα να ενημερώσω εδώ τους ευρωβουλευτές ότι η δήλωση αυτή θεωρήθηκε, μάλλον εξετάστηκε πολύ προσεκτικά και δεν ήταν τυχαία. Και είναι η καλύτερη απάντηση που μπορώ να σας δώσω για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και τις πληροφορίες. Θεωρώ πως το ζήτημα του Ιράκ είναι τραγικό αν δούμε με ποιον τρόπο εγκαταλείπουμε τώρα το Ιράκ αν μου επιτρέπετε να το διατυπώσω έτσι. Πρέπει να πω πως η εκστρατεία 2002-2012 κατέληξε σε καταστροφή. Και δεν μας τιμά καθόλου αυτό. Εντάξει, έφυγε ο αυτό είναι καλό, αλλά το τι επιτύχαμε είναι απλώς καταστροφή πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν, πόσοι άνθρωποι θα πεθάνουν ακόμα. Η χώρα έχει καταστραφεί. Οι μειονότητες είναι στην κατάσταση που είναι. Είναι απλώς καταστροφή το αποτέλεσμα αυτό, μια ανθρώπινη τραγωδία. Και σημείο καμπής στην εξασθένηση της δύση υλικής και μη υλικής. Και έχω την αίσθηση πως και στο Αφγανιστάν τα ίδια θα γίνουν. Αυτή την αίσθηση έχω. Και δυστυχώς, αν δεν προσέξουμε, έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Τώρα. για το στρατόπεδο Άσραφ και την ασφάλεια των Ιρανών εκεί πέρα. Η ασφάλεια αυτών των ανθρώπων είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως κανείς δεν μπορεί να ηγηθεί σε βάθος χρόνου στο Ιράκ. Κανείς. Ούτε η Δύση που άφησε το Ιράκ έτσι όπως το άφησε. Και ακόμη λιγότερο η Ιρακινή κυβέρνηση. Οπότε η λύση προσπαθήσουμε να μετακινήσουμε αυτούς τους ανθρώπους σε τρία βήματα, όπως ανέφερε ο κύριος Κόμπλερ, είναι ο μόνος τρόπος προστασίας αυτών των ανθρώπων. Όσο δύσκολοι και αν είναι. Στο παλιό αυτό στρατόπεδο δεν θα έχουν καμιά τύχη. Κανείς δεν τους θέλει. Και Κανείς από εμάς δεν θα τους υπερασπιστεί εκεί πέρα. Μόνο ένα τηλεγράφημα. Στείλουμε με συλληπιτήρια. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν ένα μέλλον σε διάφορες χώρες που θα τους δεχτούν. Και πρέπει να το συζητήσουμε και εμείς στις χώρες μας. Πόσους θα πάρουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να βοηθήσει εδώ πέρα η διεθνής κοινότητα. Γιατί δεν έχουμε δεν έχουν ελπίδα να πάνε στο Ιράν, αν θέλουν να επιζήσουν. Και δεν μπορεί να ξαναστηθεί όλο αυτό το στρατόπεδο εν είδη απικίας κάπου αλλού. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Κόμπλερ για τη δουλειά που κάνετε από αυτές τις δύσκολες συνθήκες τους εκπροσώπους του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ κλπ. Για να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για αυτούς τους ανθρώπους. Και εμείς ως Επιτροπή πρέπει να το ξέρουμε. Ε, εντάξει, όπως είπα εδώ πέρα, έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά το βασικότερο είναι η διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Αυτό πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Συζήτηση για την γνωμοδότηση θα γίνει 27 Μαρτίου. Γιατί δεν ήθελα να διακόψω αυτή τη συζήτηση. Αύριο το πρωί ξεκινάμε με τις ψηφοφορίες για τις εκθέσεις που ξέρετε. Εγώ δεν θα είμαι εδώ πέρα αύριο το πρωί. Πρέπει να γυαλίσω τα παπούτσια και να πάω στο Λουξεμβούργο για να συνομιλήσω με τον ε, μεγάλο δούκα του, του Λουξεμβούργου. Αυτά και σας εύχομαι καλό σας βράδυ. Und Gespräch mit dem Großkanzler Kühn, der Präsident des Europäischen